Dear colleagues, it is time to start our exchange of view with Mr. Miko, Deputy Director General for Food Safety of DG Sante, on the state of play. Θα μιλήσουμε τώρα όσον αφορά τα τρόφιμα, να δούμε πώς είναι η κατάσταση όσον αφορά τα επιστημονικά κριτήρια για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Starting our meeting, I have to πριν όμως την έναρξη της συνεδριάσεως, θα πρέπει να ευχηθούμε καλό. Όρισαν κάποιοι προσκεκλημένοι του συναδέλφου Γκίζεκε. Έτσι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην κοινωνία των πολιτών. Γι' αυτό σας έχουμε εδώ κοντά μας. Και επίση είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μας να βλέπετε εσείς πως εμείς δουλεύουμε εδώ. Και σας ευχαριστούμε για αυτό που ήρθατε. Και τώρα. Αρχίζουμε. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μίκο. Να ακούσουμε ποιες είναι θέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και στη συνέχεια, ως συνήθως, θα ακολουθήσει συζήτηση. Ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Α ξεκινήσω ευχαριστώντα σα, μου δώσατε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Να δούμε τι γίνεται όσον αφορά αυτά τα κριτήρια για του ενδοκρινικού διαταράκτε. Αυτό θα αφορά η σημερινή μου παρουσίαση. Να σα εξηγήσω ποιε είναι οι αλλαγέ στο αρχικό σχέδιο κειμένου που έχει συζητηθεί στι 18 Ενδεκάτου με εμπειρογνώμονες αλλά και κράτη-μέλη. Απλώ πρέπει να σα πω ότι για να έχουμε όσο γίνεται περισσότερη διαφάνεια Ήδη αυτό το αναθεωρημένο κείμενο έχει δημοσιευτεί στο website της Κομισιόν και τα έχουμε πει σε τεχνικό επίπεδο και με τους συνεργάτες σας. Γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι προσπάθειές σας δείχνουν εσείς πώς σημασία αποδίδεται σε όλα αυτά. Είναι η συζήτηση πολιτικού χαρακτήρα και καμιά φορά κατηγορηθήκαμε ότι δεν προστατεύουμε όσο χρειάζεται την ανθρώπινη υγεία. Όμως, σας διαβεβαιώ ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Τα προτινόμενα κριτήρια αποσκοπούν στην προστασία της υγείας όσο γίνεται καλύτερα και επομένως να έχουμε την αντίστοιχη νομοθεσία. Πρόκειται να έχουμε κριτήρια για να έχουμε καλύτερη κοινοτική πολιτική για τους διαταράκτες και αυτό γιατί τα ενδιάμεσα κριτήρια, αυτά τα οποία τώρα ισχύουν, σίγουρα δεν εξυπηρετούν τον δέοντα σκοπό, άρα πρέπει να αντικατασταθούν το γρηγορότερο δυνατόν από πιο αποτελεσματικά. Βέβαια θα πρέπει να δούμε διάφοροι ενδιαφερόμενοι τι έχουν πει, γι' αυτό και εμεί να του καλύψουμε, βελτιώσαμε το σχέδιο κειμένου, προσπαθήσαμε να το κάνουμε σαφέστερο. Πρώτα πρώτα, έχετε πει ότι αυτά τα κριτήρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. μόνο λαμβάνουν υπόψη γνωστές επιπτώσεις των διαταρακτών. Ε, και όχι ε, κάποιες επιπτώσεις που δεν έχει αποδειχθεί ότι ισχύουν. Εμείς ε, προσπαθούμε όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη και επίσης λέτε ότι ζητούμε πάρα πολύ στέρες και απαιτητικές αποδείξεις και όσον αφορά το βάρος της απόδειξης. Ναι, ναι, ναι, τα λέω πιο σιγά για να προλαβαίνουν οι διερμηνείς, λέει ο μιλητής ε, λυπούμε συνάδελφοι, θα το λάβω αυτό υπόψη. Άρα, ε, αμφισβητήθηκε το κατά πόσο είναι σωστά ρυθμίζουμε το, το βάρο απόδειξη. Αυτό δεν ισχύει. Γιατί είπαμε ότι έχουμε κάποιο είδους δεδομένα από πειράματα με ζώα και ε, αυτό περιλήφθηκε στα κριτήρια του Ιουνίου. Όμως, για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε αυτό το κείμενο είπαμε να, δια, να οι λέξεις known to cause an adverse effect και αυτού να πούμε show an adverse effect. Δηλαδή όχι είναι γνωστό ότι παράγουν αυτές τις επιπτώσεις, τις παρενέργειες, αλλά που αποδεικνύεται ότι. Οπότε έτσι θα προχωρήσουμε σε αυτή την νομοθεσία και επίσης είπαμε ότι τα καρκινογόνα είναι κατηγορία 1α. Όμως είπαμε ότι ε, εάν ε, έχουμε ε, άλλου είδους κατάταξη επί τη βάση ανθρωπίνων ενδείξεων, τότε θα πάμε στο 1B. Στο 1B είναι οι φερόμενη ως, ε, τα φερόμενα ως καρκινογόνα επί τη βάση ε, ενδείξεων από ζώα. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς δεν θα έχουμε κάποιο είδους παρερμηνία και πώς θα έχουμε τη σωστή κατάταξη στους διαταράκτες. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να υποκαταστήσουν τον κανονισμό CLP. Επίση, έχει λεχθεί ότι αυτέ, αυτά τα συμπεράσματα μπορεί να βασιστούν σε πειράματα με ζώα και όχι σε ανθρώπους. Και άρα θέλετε να έχουμε συμπεράσματα από, από ανθρώπινα, κριτήρια από ανθρώπινες έρευνες και πειράματα και αυτό και κάναμε. Ελπίζω ότι αυτό το οποίο σα ξεκαθαρίζω πρόκειται να βοηθήσει, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαριστεί ότι αυτή είναι η σωστή ερμηνεία. Επίσης, αυτά τα κριτήρια βάζουν μια καινούρια διατύπωση. Make adverse ε, effects. Ακριβώς για να καλύτερη ισχύουσα νομοθεσία. Κάναμε αυτό το οποίο ζητήσατε σε προηγούμενες επαφές μας δύναται δηλαδή να προκαλέσουν κλπ. Επίσης ζητήστε να γίνει κάποιο είδους εντοπισμός και αυτός να γίνεται μόνο επί τη βάση κάποιων μελετών που γίνονται σύμφωνα με κάποιο είδους διεθνή και αποδεκτά πρωτόκολλα. Δηλαδή υπήρχε ο φόβος ότι κάποιες από τις μελέτες πρόκειται να μην ληφθούν υπόψη από την αξιολόγηση και για να μπορέσουμε να σας καλύψουμε, το εφηρημένο κείμενο διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει κάποιο είδους ε, ιεραρχία όσον αφορά το τι είδους επιστημονική τεκμηρίωση θα ληφθεί υπόψη για τον εντοπισμό των ε, διατρακτών. Όμως εμείς έχουμε την ίδια δομή όπως και προηγουμένως όσον αφορά του είδους βιβλιογραφία θα μελετήσουμε. Ακριβώς όπως συνιστούν οι επιστήμονες. Η γενικότερη προσέγγισή μας σε αυτά τα κριτήρια του Ιουνίου δεν έχει μεταβληθεί. Τα αναφερμένα κριτήρια δεν καλύπτουν κάποιες κατηγορίες που δεν είναι επιθυμητό. Ούτε θέλουμε μεταβατική περίοδο. Θέλουμε αυτά τα κριτήρια να ισχύσουν με την θέση σε ισχύ του κειμένου. Όσον αφορά τώρα αυτή την ε, τροπολογία για την παρέκκληση, δεν θα αλλάξει τίποτα. Ξέρω ότι εσάς αυτό σας ανησυχεί. Η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου έχει γνωμοδοτήσει και συμπεραίνει ότι εδώ υπάρχει υπερβάση γνωμοδοτήτων από την Κομισιόν. Γνωρίζω δε τι έχουν πει. Αλλά σας ε, επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπε ε, προς τον κύριο Λαβία, προς την Επιτροπή σας, ο Αρμόδιος Είμαστε πεπισμένοι ότι το άρθρο 78 αυτού του είδου του κανονισμού για την προστασία των φυτών δίνει στην ε, Κομισιόν την αρμοδιότητα να τροποποιήσει τις ε, τεχνικές λεπτομέρειε λαμβάνοντα υπόψη την ισχύουσα τεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση και οι βασικές ε, παρεκκλήσει όσον αφορά κάποιο είδου αμεληταία έκθεση έχουν να κάνουν με κάποιο είδου επίση αμεληταίου κινδύνου από αυτή την έκθεση ή την έκθεση σε αυτούς τους παράγοντες. Αυτό είναι επιστημονικό και σας παραπέμπουμε γενικότερα στους επιστήμονες και στις, ε, και στις δημοσιεύσεις ε, της, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Διατροφική Ασφάλεια του 2013 και άλλων το 2014. Επίσης, λέμε σε αυτή την ε, τροπολογία ότι οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε δεν θεωρηθεί ότι είναι διαταράκτες, ό,τι δηλαδή δεν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, δεν θεωρείται διαταράκτες. δεν εγκρίνεται. Έτσι θεωρούμε ότι κάνουμε ό,τι λέει η επιστήμη. Έτσι επίσης εξασφαλίζουμε την προστασία της υγείας. Δηλαδή, έτσι εξασφαλίζουμε ότι κάποιες επικίνδυνες ουσίες δεν θα εγκριθούν σύμφωνα με την παρέκκληση, ακόμα και αν έχουμε έκθεση αμεληταία. Όπως σας προείπα, αυτές οι αλλαγές συζητήθηκαν με τα κράτη-μέλη και τους συμπεριγνώμενε στις 18 Νοεμβρίου και σας πληροφορώ ότι πάρα πολλές αντιπροσωπείε κρατών μελών ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί επίσημα για τα κριτήρια. Παρά τι προσπαθίε μα να καλύψουμε κάποιες ε, ανησυχίε, κάποια κράτη ακόμα θέλουν να γίνει και άλλη αναθεώρηση του κειμένου. Κάποια άλλα κράτη συμφωνούν το κείμενο όσο έχει τώρα. Γι' αυτό τα κράτη-μέλη είπαν ότι θα πρέπει να υποβληθούν οι παρατηρήσεις μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Αύριο δηλαδή. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε τι άλλες αλλαγές θα γίνουν τόσο ώστε να ε, καλύψουμε τις παρατηρήσεις των κρατών μελών και όπως γνωρίζετε εάν δεν υπάρξει συμφωνία για κάποιο είδους, για κάποιο συμφωνία λογική, ε, τότε θα συνεχίσουν να ισχύουν τα σημερινά ισχύουν κριτήρια ακόμη και αν εξυπηρετούν τον τεθέντα σκοπό όπως λένε όλοι. Δεν θα υπάρξει σωστή επισήμανση των διατρακτών. Θα πρέπει να γίνει αλλαγή το συντομότερο δυνατόν. Γι' αυτό εμείς υπολογίζουμε στην δική σας υποστήριξη, ούτως ώστε το ταχύτερο να αποφασιστεί ό,τι καλύτερο για τα κριτήρια αυτά. Τελευταίο που έχω να σας πω είναι το ότι στο μεταξύ, για να μην χάνουμε χρόνο, από την ΕΦΣΑ και την ΕΓΑ, να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα έγγραφα τα σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων. Και έτσι να έχουμε άμεση ισχύ τους όταν τεθεί το νομοθέτημα σε ισχύ. Όλα αυτά τα οποία ήδη έχουν ανέβει και δημοσιευτεί στο website. Αυτά και περιμένω την αντιδράσή σας, τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκίζεγε είναι ο πρώτος που θα κάνει ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Μίκο, να πληρωτή διευθυντή, όσον αφορά την πρόταση της ε, Επιτροπής και μετά τη θέσπιση επιστημονικών δεδομένων και κριτηρίων Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι για να εγγυηθεί και να προστατεύσει την υγεία μας παραμένει μέσα στον ανταγωνισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πολύ καλή πρόταση αυτή που μας υποβάλλει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα κάνω λοιπόν και τρία σχόλια, τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, το θέμα της δόσης είναι πολύ σημαντικό. Η δόση είναι αυτή που κάνει κάποια ουσία δηλητήριο και επικίνδυνη. Υπάρχουν λοιπόν ουσίες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν στην ε, φύση, να μην ε, πλήττουν σε μικρές δόσεις, να μην είναι επιβλαβείς, αλλά σε μεγαλύτερη δόση ή μεσισόρευση να είναι θανατηφόρες. Οι ορμονικοί διαταράκτες λοιπόν, και αυτή είναι η συσσόρευση, να ειναι θανατηφορες οι ορμονικοι διαταρακτες παρατήρησή μου, θα πρέπει να μπουν σε σωστές κατηγορίες είναι κάτι που σίγουρα μπορεί να δημιουργήσει πολύ σημαντικές ανισορροπίες και στρεβλώσεις και όσον αφορά τη χρήση των ε, παρασιτοκτόνων. Αλλά είναι πολύ σημαντικό οι άδειε που δίνονται και οι επιπτώσεις στη βιομηχανία να υπολογιστούν σωστά. Τρίτον, οι λεγόμενοι κίνδυνοι, δευτερεύοντες κίνδυνοι, και οι σημερινές ρυθμίσεις και κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να προσαρμοστούν στα πολύ πρόσφατα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σήμερα σίγουρα θα πρέπει να δημιουργήσουμε κανόνες και ρυθμίσεις οι οποίοι να είναι συμβατοί και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό ε, Εμπορίου και οι αναλύσεις της Επιτροπής αλλά και η ΕΦΣΑ θα ενσωματώσουν και πρέπει να ενσωματώσουν όλες αυτές τις προϋποθέσεις και τα στοιχεία και είναι πολύ σημαντικό σήμερα να λάβουμε υπόψη μας και να αποτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε σωστά τους κινδύνους βάσει των νέων επιστημονικών δεδομένων. Δεύτερον, το θέμα της, του ανταγωνισμού, της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και του εμπορίου. Λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει λοιπόν να επεξεργαστεί εκ νέου όλα αυτά τα δεδομένα που την οδηγούν στη θέσπιση των προδιαγραφών. Ο κύριος Μίκο το είπε πάρα πολύ σωστά. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καθυστερήσουμε και να αναβάλουμε. Χρειαζόμαστε νομική ασφάλεια για όλους τους εμπλεκόμενους ε, σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πότς. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα απ' όλα που πάει κάπως προς τη δικιά μας κατεύθυνση. Όμως λίγο πλησιάζει προς αυτό το οποίο χρειάζεται. χρειάζεται ακόμα πιο διαφορετική προσέγγιση. Κυρίως και πρώτα απ' όλα γιατί τα κριτήρια πρέπει να είναι οριζόντια και να εφαρμόζονται σε άλλους κανονισμούς κλπ. και Αυτά είναι στα λόγια. Υπάρχουν κριτήρια για ένα τμήμα της νομοθεσίας και αυτό είναι και η αδυναμία όλων των προτάσεων. Και έπειτα και πρακτικές παρατηρήσεις. Μιλήσατε για μετρήσιμο κινδύνο, κίνδυνο και έκθεση. Ακόμα και αν δεχτώ τα επιχειρήματα που μας παρουσιάσατε, αν θυμάμαι καλά το κείμενο της πρότασης, η Επιτροπή το χρησιμοποιεί αυτό μόνο για τις εξαιρέσεις. Μόνο σε άλλα σημεία του κειμένου χρησιμοποιείται την ε, διατύπωση για την ε, ασήμαντη έκθεση δηλαδή στην περίπτωση ενός ε, μιας ουσίας ακολουθείται διαφορετική προσέγγιση βάσει εξαιρέσεων και σε άλλη περίπτωση βάσει κινδύνου. Οπότε ρωτάω, Γιατί υπάρχει αυτή η αλλαγή, μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Όσον αφορά τους ορισμούς, και εδώ έρχομαι στη δεύτερη ερώτησή μου, η Επιτροπή πάντα έλεγε ότι πρέπει να βασιστούμε στους ορισμούς της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Πάντα το λέει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως φοβάμαι ότι αν δούμε το 36522 της πρότασης, αναγνωρίζει η Επιτροπή το γεγονός και σύμφωνα με τον ΠΟΗ θα πρέπει να λέει όπου υπάρχει πόνοια ότι προκαλεί βλάβη. Έχει κάνει αλλαγές δηλαδή η Επιτροπή στη διατύπωση του ΠΟΗ αλλάζει το σύστημα ενδοκρινικών διαταρακτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά δεν βασίζεται στον ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Οπότε ρωτάω, οι αλλαγές που επιφέρετε, της Κομισιόν βέβαια, εντάξει όχι προσωπικά του κ. Μίκου, προφανώς, δεν μπορεί να παραμείνουν κάποιοι επικίνδυνοι διαταράκτες εκτός πεδίου εφαρμογής του κειμένου αυτού, εξαιτίας ακριβώς των αλλαγών που έχετε επιφέρει στους ορισμούς ε, της ΠΟΗ. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Γκέρλινγκ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μίκο που ήρθε σήμερα. Θέλω να επαναλάβω και εγώ τα σχόλια που κάναμε εδώ στην Επιτροπή μας και τον Ιούνιο. Δεν ήμουν έτσι κι αλλιώς 100% ευχαριστημένη από το σχέδιο που είχαμε. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Απογοητεύομαι επειδή επέλεξε την επιλογή 2 και όχι την 4 η Κομισιόν. Ξέρω ότι στις αρχικές αντιδράσεις ήμουν μειοψηφία, οπότε δεν περίμενα ότι θα το έχει αλλάξει αυτό. Αλλά, βάση περιπτώσει, ήλπιζα ότι θα φτάσουμε σε κάποιο συμβιβασμό. Να έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία να μας ικανοποιούν όλους. Λοιπόν, για να σχολιάσω τώρα συγκεκριμένα στις αλλαγές που έχουν γίνει. Σημειώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει προσπάθειες να ευθυγραμμίσει τους ορισμούς της με εκείνους ε, της ΠΟΗ. Ήτανε ένας από τους ε, με τις βασικές επικρίσεις που είχαμε στην αρχή. Αλλά βέβαια ότι και τώρα είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι. Χαίρομαι πάντως ότι αποσαφήνισε κάπως το κείμενο που δεν ήταν τόσο μπερδεμένο που αναφερόταν σε δοκιμές τους ανθρώπους και είχαν ακουστεί πολλά από αυτούς στην τελευταία συνάντηση. Επίσης αντιστάθηκε στο να δημιουργήσει κατηγορίες. Δεν ήταν βέβαια αυτό που προτιμούσα, Χαίρομαι επίσης που αντιστάθηκε η Επιτροπή στο να βγάλει τις τροποποίησεις όσον αφορά τις εξαιρέσεις. Ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνούν, αλλά εγώ πιστεύω ότι η προσέγγιση βάση κινδύνου είναι η πιο αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Για μένα αυτό υπερισχύει. Τέλος, υπενθυμίζω ότι αν απορρίψουμε αυτό το κείμενο, επιστρέφουμε στα προσωρινά κριτήρια, τα οποία δεν ικανοποιούσαν κανένα. Εδώ έχουμε μπροστά μας μια σημαντική βελτίωση όσον αφορά τα προσωρινά κριτήρια και με ένα συμβιβασμό νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπή πια και μπορούμε και εμείς να προχωρήσουμε και να μην παραμείνουμε κολλημένοι να τελειώσει πια αυτή η αβεβαιότητα που υπάρχει και να εγκριθούν τα κριτήρια. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριο Εικάουτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον κύριο Μίκο που ήρθε και μας έδωσε αυτές τις εξηγήσει. Θέλω να αρχίσω με το σχόλιο του κύριου Μίκο που είπε ότι έχει πολιτικοποιηθεί πολύ αυτή η υπόθεση. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τελικά ποιος το πολιτικοποίησε. Και εδώ μία πλευρά πολιτικοποίησε από την αρχή αυτό το ζήτημα και αυτή ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μπήκε σε μία αξιολόγηση οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων ήδη από το 2013, όταν είχαμε πει όχι, μην το κάνετε και όχι με αυτόν τον τρόπο. Συνέχισαν όμως, οπότε ακόμα και το δικαστήριο χρειάστηκε. Και ακόμα και αφού είπε το δικαστήριο Ευρωπαϊκή πρέπει να έρθετε με επιστημονικά κριτήρια και σταματήστε με την ε, αξιολόγηση αντικτύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέχισε. Και το λέω και προ τη συνάδελφο την κυρία Γκέρλινγκ, ότι είναι το ρυθμιστικό συμβούλιο το οποίο ήρθε τον Ιούνιο. εμεί ποτέ δεν θέλαμε αυτό το ε, ρυθμιστικό εποπτικό συμβούλιο. Η Τζούλη Γκέρλινγκ πίεζε γι' αυτό. Τι είπε? Είπε ότι ότι δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε μία ουσία βάσει υποθέσεων και ότι πρέπει να υπάρχει σωστή αξιολόγηση. Και είπε επίση ότι η σημερινή αξιολόγηση δεν είναι αντικειμενική. Αυτά είναι πολύ σκληρά λόγια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν τα λέμε εμείς, τα λέει το Συμβούλιο αυτό το εποπτικό ρυθμιστικό. Οπότε άμα λέτε εσεί ότι πολιτικοποιήθηκε, ε, για κοιτάξτε ποιο το πολιτικοποίησε πρώτα απ' όλα. Καταλήξαμε στα δικαστήρια γι' αυτό το λόγο. Ε, καλό θα ήταν να έχουμε και λίγη αυτογνωσία όταν μιλάμε. Τώρα πού βρισκόμαστε. Ξέροντας ότι ήθελε την επιλογή 4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ήθελε να πάει εκεί, απογορεύτηκε. Σας είπαν δεν γίνεται, δεν μπορείτε. Οπότε έπρεπε η Επιτροπή να βρει κάποια άλλη λύση. Και ήμασταν επικριτικοί για δύο λόγους. Πρώτον όσον αφορά τα κριτήρια και δεύτερον όσον αφορά την τροποποίηση στην εξαίρεση. Αυτά τα δύο τμήματα μας ενοχλούσαν και εξακολουθούν να μας ενοχλούν. Δεν μου αρέσει να είμαι επικριτικό, αλλά δεν έχουν αντιμετωπιστεί κάποια ζητήματα, δεν έχουν λυθεί και για να σας βάλω κάποια ερωτήματα. Κοιτάξτε, είναι ίσως το πιο σημαντικό αυτό. Πρόκειται για τις τρεις εντολές που αλλάζετε, όμως εξακολουθείτε στο σημείο 2 να έχετε τον ορισμό της ενδοκρινικής δράσης. Δεν είναι όμως αυτός ο ορισμός της ΠΟΕ, που είναι ότι τροποποιεί τη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από τον ενδοκρινικό τρόπο δράσης. Γιατί χρησιμοποιείται μια διαφορετική διατύπωση λοιπόν από την ΠΟΕ, γιατί ρωτάω. Δεύτερον, πού Έπειτα, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται να ακολουθήσει τις διαδικασίες του ΣΠΟΕ και οι αυτέ αυτές τις τρεις εντολές. Και κάτι προς την Ζούλη Γκάρλινγκ πάλι. Ξέρω ότι τοποθετήσετε πολιτικά. Εδώ όμως συζητάμε και ένα νομικό ζήτημα και την θέση του συνομοθέτη. Όταν λοιπόν τον Ιούνιο είχαμε επικρίσεις ζητήσαμε να το κοιτάξουν και οι νομικές υπηρεσίες. Οπότε, πρώτα το δικαστήριο, μετά το συμβούλιο το ελεγκτικό και μετά είχαμε και πολιτική αντίδραση ότι δεν τα κάνει καλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εξακολουθεί στον ίδιο δρόμο. Η Επιτροπή βέβαια μας απάντησε, απάντησε στο Κοινοβούλιο λέγοντας «Μα όχι, η αλλαγή στην προσέγγιση βάση κινδύνου είναι για καλύτερη προστασία. Δηλαδή προσπαθεί να μας πείσει ότι το κάνει για μας. Ναι, αλλά αλλάζει ένα νομικό στοιχείο. Και λέει ότι το κάνει για μας, που είμαστε εμείς οι συνομοθέτες. Και έχω εδώ τώρα το νομικό έγγραφο, τον Ιούλιο. Η Επιτροπή μίλησε και με κάποιους πρέσβεις Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και άλλων χωρών οι οποίοι πιέζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνει την προσέγγιση αυτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει, μα ξέρετε, εμείς πρέπει να έχουμε την προσέγγιση βάσει της βλάβης, αλλά τελικά κάποιος είπε, για κοιτάξτε την πρόταση που προβλέπει τη δυνατότητα να επανέλθουμε σε αυτά τα επίπεδα ουσίας. Και εσείς προσπαθείτε να μας πείτε ότι καθησυχάσετε με αυτόν τον τρόπο τις ανησυχίες μας. Δηλαδή εσείς μας λέτε σας δίνουμε περισσότερη προστασία, ενώ συγχρόνως τους πρέσβει τη Ουρουάη, των ΗΠΑ, του Καναδά κτλ. τους πουλάτε το ότι τι δικέ του ανησυχίε ε, καθησυχάζετε για τη διαφορετική προσέγγιση. Μα δεν μπορείτε να τάξετε και τα δύο. Και το έγγραφο αυτό ακριβώς δείχνει τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αλλάζει την νομοθεσία γιατί πιέζεται από διεθνείς παράγοντες και ο στόχος της είναι να αλλάξει το νόμο. Λοιπόν, Τζούλι Γκέρλινγκ, να το ξέρεις αυτό. Αν θέλουν να το κάνουν, να το κάνουν με την σωστή νομοθετική διαδικασία και όχι με αυτόν τον τρόπο δράσης. Γιατί το έχουν ήδη εξηγήσει οι νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και ισχύει. Λοιπόν, λυπάμαι, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι, έχει πολιτικοποιηθεί πολύ το θέμα, αλλά εσείς το πολιτικοποίησατε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, επεξηγήσεις. Υπενθυμίζω ότι η Επιτροπή πρότεινε κάποια κριτήρια για τους ε, διαταράκτες μετά την προθεσμία που προβλεπόταν για από τα διοκτώνα και από τα ε, παρασιτοκτώνα στους κανονισμούς και πολύ αργότερα από ε, τα όσα είχε κρίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπότε είδαμε ότι στο τσακ γλίτωσε τότε και την ε, πρόταση της πιστείας. Τώρα έχουμε κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Ακόμα και αυτές τις τόσο ελαφρές τροποποιήσεις τις επικρίνουν τα κράτη-μέλη. Επομένως για τους διαταράκτες τι ξέρουμε Ξέρουμε τι είπε ο Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ότι θα πρέπει να απαγορευτούν ακόμα και εκείνες οι ουσίες που δύναται να παράξουν τα ίδια αποτελέσματα. Και είπαμε ότι αν είμαστε προσεκτικοί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις παρεκκλήσεις. Άρα χρειάζεται να υπάρχει αρχή της σοφροσύνης. Προσοχή στις τροπολογίες και στις διαπραγματεύσεις, τι θα προκύψει με Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Υπάρχουν τώρα οι κλάδοι που ενδιαφέρονται, όπως με τα διοκτώνα, όπως με τα ζανιοκτώτα. Αν όμως περάσει αυτή η πρόταση, θα έχουμε ε, αυτές τις ουσίες παντού, σε φάρμακα, σε, σε καλλιντικά, σε τρόφιμα. Άρα τα πράγματα θα έχουν και τώρα, δεν θα βελτιωθεί τίποτα. Επομένω, δεν λαμβάνετε τίποτα απόψε από τις εξελίξεις που έχουμε γύρω-γύρω. Κύριε Αντόρνονα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθυντά, το θέμα των ε, νομικών διαταρακτών είναι στην επικαιρότητα. Εκατό επιστήμονες ε, δημοσιεύουν σήμερα ένα άρθρο στην εφημερίδα Le Monde που αφορά την δράση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία πραγματικά δεν αναφέρει την επικινδυνότητα αυτών των ουσιών στο πραγματικό της επίπεδο. Τι χρειάζεται για να αντιδράσουμε καρκίνη του μαστού των γεννητικών οργάνων, καθώς και άλλες πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία που σήμερα αποδεικνύονται από τους επιστήμονες είναι αποδεδειγμένοι πλέον και αυτό που σήμερα μας απασχολεί είναι τι είναι και τι δεν είναι ορμονικός διακταράκτης. Πιστεύω ότι καλύτερα θα κάνουμε να ασχοληθούμε εμείς και η Επιτροπή με την αρχή της προφύλαξης κάτι το εξαιρετικά επίγον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να δεσμευθεί για την προστασία της ε, δημόσιας υγείας των Ευρωπαίων πολιτών και να σταματήσει να στηρίζει τα βιομηχανικά και οικονομικά συμφέροντα των ε, ευρωπαϊκών εταιριών. Γίνεται μια πολύ συγκεκριμένη έκκληση και αναρωτιέμαι αν πραγματικά οι ελεύθερες συναλλαγές και το ελεύθερο εμπόριο προέχει ενός αποτελεσματικού ελέγχου για τους ορμονικούς διαταράκτες. Ξέρετε ποια είναι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν επιθυμούν περιορισμού στη χρήση αυτών των ουσιών. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να περιμένουμε την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά την αυστηρότητα της νομοθεσίας μας. Αν ναι, τότε κατανοούμε γιατί δεν υπάρχει δράση σε αυτό το τομέα. Μία δράση που είναι απαραίτητη. Ξέρω ότι υπάρχουν και εσωτερικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αμφισβητούν τις ε, πληροφορίες και τα στοιχεία της ΕΦΣΑ, θεωρώντας αυτές τις δηλώσεις μεροληπτικές και όχι επιστημονικά αποδεδειγμένες. Ε, μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε αυτές τις δηλώσεις σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντάλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστούμε για την Επιτροπή που ήρθε, μας τα διευκρίνησε και μας παρουσίασε τη θέση τους, Μας απαντά και τις ερωτήσεις. Πάντως το θέμα είναι ότι αυτή η πρόταση δεν είναι ρεαλιστική όσον αφορά το τι αποδείξεις και ενδείξεις επιστημονικές θέλει για την επισήμανση των διατρακτών και την έγκριση αυτών και σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε αρνητικές επιπτώσεις από χημικές ουσίες γιατί υπάρχουν δεδομένα που κατατείνουν στο να αποδείξουν αυτό και βλέπουμε πως διαταράσσεται το ενδοκρινικό σύστημα και ότι από τους διαταράκτες προκύπτει αυτό το αποτέλεσμα αλλά η απόδειξη είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει άρα θα πρέπει να δούμε πως θα ανοιχνεύεται αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα να δούμε πώς θα υπάρχει η απόδειξη της σχέσης αιτίου και αιτιατού. Άρα Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα τάσει πάρα πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, βάζει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη για την απόδειξη που απαιτείται. Και ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε αυτή η η αλλαγή όσον αφορά το αν επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα ζενιοκτόνο εάν ε, έχουμε αμελητές επιπτώσεις. Όμως έχει συμφωνήσει με τη συναπόφαση και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ότι ο κανονισμός προστασίας των φωτών, των φυτών ε, ήταν κάτι στο οποίο συμφωνήσαν και τα τρία θεσμικά όργανα και είπαμε ότι εκεί είχαμε εφαρμόσει αρχή της προφύλαξης. Άρα γιατί θέλει να το αλλάξει αυτό όσον αφορά την έκθεση των καταναλωτών. Τέλος. Βέβαια στον όσο ακούσαμε από την Επιτροπή. Εάν έχουμε ειδική πλειοψηφία η οποία δεν προκύψει σε επίπεδο τεχνικής επιτροπής, το RPS προβλέπει ότι μπορούν οι υπουργοί σε πολιτικό επίπεδο στο Συμβούλιο να αποφασίσουν. Θα το κάνει αυτό η Επιτροπή και να αποφασίσουν επομένως στο Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Μίκο που είναι σήμερα εδώ. Εγώ θα μιλήσω για το σύριαλ των ε, ορμονικών διαταρακτών. Εδώ και τόσα καιρό ξεκινήσατε με τη θέσπιση προτύπων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφανθεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο και τώρα ξαφνικά βλέπουμε κάποιες προτάσεις με τις οποίες συμφωνούν οι περισσότεροι. Εάν η Επιτροπή όμως δεν παίξει το ρόλο του θεματοφύλακα της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών καταλαβαίνετε ποιο θα είναι ο αντίκτυπος των Ευρωπαίων πολιτών επί των Ευρωπαϊκών θεσμών. Υπάρχει, όπως ξέρετε, μια αναφορά με χιλιάδες υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε την Endocrine Society με χιλιάδες ε, επιστήμονες που αμφισβητούν τα κριτήριά σας. Πείτε μου τι άλλο θέλετε για να αντιδράσετε. Έχουμε την επιρροή από μέρους των Καναδών, των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαβάστε και την εφημερίδα Le Monde που αναφέρεται στην ΕΦΣΑ και στα πορίσματά της από το Δεκέμβριο του 2012. Η περίφημη ΕΦΣΑ με τις ε, μελέτες της, που δεν μπορούν βεβαίως να μας τις δημοσιεύσουν, που αναφέρεται στους ορμονικούς διαταράκτες λέγοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως και όλα τα άλλα επικίνδυνα για την υγεία προϊόντα. Κύριε Μίκο, συμφωνείτε με αυτόν τον ορισμό. Γιατί όταν κοιτάξει κανείς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, διαφωνεί με αυτόν τον ορισμό. Αναφέρουν την παραδοσιακή μέθοδο αξιολόγησης για τα χημικά προϊόντα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να ισχύει για την περίπτωση των ορμονικών διαταρακτών. Αναρωτιέμαι λοιπόν και επειδή καταλήγουν σε διαφορετικό συμπέρασμα από εσά, αν συμφωνείτε ναι ή όχι με αυτήν την διαπίστωση. Το θέμα τώρα του κινδύνου και της έκθεσης του ανθρώπου σε αυτές τις ουσίες. Η λογική της Επιτροπής είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, διότι περνάτε από την αξιολόγηση του κινδύνου στην αξιολόγηση του ρίσκου. Δηλαδή, προσπαθείτε να μην λάβετε υπόψη σας αυτό που ο νομοθέτης θέλησε, θέλησε να συμπεριλάβει στα κείμενα. Προσπαθείτε να παρεκκλίνετε και να παρακάμψετε το εμπόδιο. Οι νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου μας είπαν ότι είναι παράνομη αυτή η μέθοδος. Όσον αφορά τώρα τα κριτήρια της Επιτροπής για τον ορισμό που επίσης δεν λαμβάνει υπόψη του την αρχή της προφύλαξης. Εγώ είμαι βιολόγος. Μου λέτε λοιπόν ότι πρέπει να αποδείξουμε τη δράση των ορμονικών διαταρακτών. Μα κοιτάξτε, εδώ έχουμε την δράση και κατόπιν τα αποτελέσματα. Είναι κάτι που θα έρθει πολύ αργότερα. Εσείς λοιπόν με τα πολύ αυστηρά κριτήρια που έχετε θεσπίσει δεν επιτρέπετε να φτάσουμε ποτέ στο αποτέλεσμα ανησυχώ πάρα πολύ. Πρώτον, για την εικόνα της Ευρώπης, για την προστασία της δημόσιας υγείας. Όταν κάποιος διαπιστώσει τι βλάβες προκαλούν στη γονιμότητα, επί της υγείας, με τους καρκίνους, στην υγεία των παιδιών. Τι άλλο περιμένετε, τι άλλο περιμένετε. Σταματήστε να στηρίζετε τη βιομηχανία όπως το κάνατε και με τον καπνό. Τι περιμένετε ακόμα για να αντιδράσετε. I uh, Καλώς. Τώρα, κύριε Μίκο, πολλές ερωτήσεις. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ όλους για τις αντιδράσεις σας και τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες και ελπίζω να μην ξεχάσω τίποτα. Πρώτον, νομίζω ότι εν μέρει τουλάχιστον εκτιμήθηκε ότι οι αλλαγές που σας παρουσίασα σήμερα αντιμετωπίζουν ζητήματα τα οποία είχαν τεθεί κατά το παρελθόν. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο ξεκάθαρος από ό,τι όταν τα παρουσίασα στην αρχή. Πρώτον, η ερώτησή σας για αυτό που θεωρήσατε βασικό, ότι δηλαδή τα κριτήρια εφαρμόζονται μόνο σε δύο νομοθετήματα και όχι σε όλα. Η απάντηση είναι απλή. Καταλαβαίνω βέβαια την λογική. Η εντολή μας όμως ήταν μόνο για τους δύο συγκεκριμένους κανονισμούς που έχουν να κάνουν με τα βιογειονομικά κλπ. Εμείς λοιπόν υποθέτουμε και πιστεύουμε ότι άπαξ και υπάρχει πολιτική συμφωνία. Έχουμε έναν ορισμό και έχουμε έναν ορισμό βάσει του συστήματος, τότε θα τροφοδοτηθεί η συζήτηση για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και στα υπόλοιπα νομοθετήματα. Αλλά η δικιά μας εντολή δεν ήταν αυτή, δεν ήταν για να ασχοληθούμε και με όλα τα άλλα. Επιπλέον πρέπει να πω ότι είναι μια αρκετά πλήρης δουλειά αυτή που χρειάζεται και πολύ περισσότερο χρόνο. Εσείς το είπατε πολλές φορές ότι φοβόσαστε ότι η παρουσία, μάλλον προστασία ε, στα φυτά και στα φυτογειονομικά ήταν το πιο σημαντικό. Και αυτή ήταν η νομική μας υποχρέωση. Τώρα άκουσα επίσης να λέτε ότι δεν αντικατοπτρίζεται ε, στις, ε, στη νέα εκδοχή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εγώ όμως θα ήθελα να σας ζητήσω να μην ερμηνεύουμε στραβά την απόφαση του δικαστηρίου, γιατί το δικαστήριο δεν είπε ότι το πρόβλημα είναι η αξιολόγηση αντικτύπου το δικαστήριο είπε ότι έπρεπε να είχε γίνει έγκαιρα. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν κακή αξιολόγηση αντικτύπη ότι δεν έπρεπε να γίνει, ότι δεν την κάναμε έγκαιρα. Αυτή ήταν η κριτική του δικαστηρίου. Και το έχω πει πολλές φορές και σε προηγούμενες συζητήσεις, δεν έχει να κάνει τόσο με τη σύνδεση με τον ε, ορισμό αλλά με την ευθύνη. Δηλαδή, αν αρχίσει να λειτουργεί ο ορισμός από την, ημέρα, την πρώτη μέρα, θα πρέπει να ξέρετε συγκεκριμένα τι θα συμβεί στο σύστημα και να είσαστε έτοιμοι γι' αυτό. Και νομίζω ότι είναι υπεύθυνο αν κοιτάξουμε τη μελέτη αντικτύπου. Η προτινόμενη πρόταση βασίζεται στην ζημιά και όχι στον κίνδυνο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες στη μία και στην άλλη περίπτωση. Τώρα για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Πολλές φορές αναφέρθηκε από πολλούς το θέμα του κινδύνου και της ε, έκθεσης. το μελιτέο κινδύνου και της αμελιτέας έκθεσης. Η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει την άποψη ότι εμείς ξεπεράσαμε τις εξουσίες μας. Όμως εμείς κάναμε την ίδια ανάλυση από τις δικές μας νομικές υπηρεσίες, ευρωπαϊκές επιτροπές που μας επιβεβαίωσαν ότι είμαστε μέσα στα πλαίσια της εντολής που μας δίνεται βάσει του άρθρου 78, όπου έχουμε αυτήν την αρμοδιότητα και να ευθυγραμμιζόμαστε με τις τελευταίες εξελίξεις, τις επιστημονικές, ορισμών κλπ. Επιμένουμε λοιπόν ότι είμαστε μέσα στα πλαίσια της εντολής μας. Βέβαια ε, μπορεί μεταξύ μας να διαφωνήσουμε ε, και δεν θα καθίσω εγώ να σας πω τώρα ποια από τις δύο νομικές υπηρεσίες είναι καλύτερη αλλά σας λέω ότι εμείς ακολουθήσαμε τη δικιά μας νομική υπηρεσία, γιατί αυτό τους ρωτήσαμε στην αρχή. Και η απάντησή τους ήταν ξεκάθαρη. Βάσει αυτή τη νομική ανάλυση, λοιπόν, τη νομική μα υπηρεσία λειτουργούμε. Αυτά για τη νομική πτυχή. Τώρα για το περιεχόμενο. Δεν μου αρέσει να μπερδεύουμε τις ερμηνείε. Στην αρχή τη συζήτηση ήταν μια πολύ δύσκολη ε, συζήτηση από τη μια πλευρά θέλαμε την πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονη προσέγγιση και από την άλλη μεριά υπήρχε πίεση και εμείς την καταλαβαίνουμε αυτή την πίεση ότι όταν μιλάμε για ενδοκρινική συμπεριφορά έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένα μόρια και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλουμε όρια. Και γι' αυτό το προτιμότερο να πάμε σε αυτό που λέμε hazard base, βάση βλάβης δηλαδή. Και αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε. Και επιμένω και το επαναλαμβάνω ότι ο ορισμός αυτός είναι hazard base. Τώρα, εκεί που εμφανίζεται ο κίνδυνος, risk, είναι σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις εξαιρέσεων. Τώρα μπορείτε να ρωτήσετε ε, θα έχουμε τέτοιες εξαιρέσεις. Μια μικρή αναλογία, δεν ξέρω πόσες θα είναι ακριβώς αυτές. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν μιλάμε για εξαίρεση πρέπει να έχουμε κάτι το οποίο θα λειτουργεί, θα είναι μετρήσιμο και που θα μπορούμε να το ορίσουμε. Οπότε σας ρωτάω, ας πούμε, αμελητή έκθεση, τι σημαίνει. Εγώ ξέρω πολύ καλά, είμαι σε θέση, έχουμε τη μεθοδολογία να ορίσουμε τι είναι αμελητέος κίνδυνος. Αμελητέα έκθεση είναι πιο ασαφής όρος. Η αμελητέα έκθεση λοιπόν σημαίνει ότι έρχεστε σε επαφή με μια πολύ χαμηλή ποσότητα της ουσίας. Έτσι φαντάζομαι με αυτό θα συμφωνήσουν όλοι. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι στην περίπτωση των ενδοκρινικών διαταρακτών ο κίνδυνος μπορεί να είναι υψηλός ακόμα και αν έρθετε σε επαφή με αμελητέα ποσότητα της ουσίας. Μπορεί δηλαδή να βρεθούμε σε καταστάσεις όπου ο αμεληταίο κίνδυνος είναι χαμηλότερος από την αμεληταία έκθεση. Και αυτό μπορεί να ισχύσει και από τις δύο πλευρές. Δεν το αρνούμε. Απλώς το ξεκαθαρίζω. Εμείς λοιπόν είμαστε πιο συγκεκριμένοι αν μιλάμε για αμεληταίο κίνδυνο και πρέπει να αποδειχτεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση κλπ. Και, και όλους αυτούς τους κανόνες που πολύ καλά γνωρίζετε. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι δεν είναι σωστό αυτό να το σαν μια αλλαγή στην προσέγγιση, γιατί ο ορισμός παραμένει hazard base. Η προσέγγιση βάσει του αμεληταίου κινδύνου είναι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μπορεί να εφαρμοστεί σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και πολύ συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Οι επικρίσεις που έρχονται τώρα από διάφορες πλευρές και από μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλους λένε Μα εμεί φοβούμαστε ότι με την προσέγγιση αυτή παρακάμπτεται τον ορισμό σας ε, βάση βλάβης και δεν θα υπάρχει καμία ουσία τελικά στον κατάλογο γιατί θα χρησιμοποιήσετε όλες τις εξαιρέσεις βάση κινδύνου. Ξαναλέω αυτό που έχω ξαναπεί βάσει των πληροφοριών που έχουμε είμαι πεπισμένος ότι δεν υπάρχει κενός κατάλογος ενδοκρινικών ε, διαταρακτών μετά από τον ορισμό αυτό. Θα είναι ένας πλήρης κατάλογος ο οποίος θα βασίζεται στον ορισμό και δεν θα είναι εύκολο να πετύχει κανείς εξαιρέσεις. Και κάτι σχετικά με αυτό. Το θέμα των MRL. Εμείς εξορισμού λέμε εάν η ουσία απαγορεύεται γιατί είναι ενδοκρινικός διαταράχτης βάσει του προτινούμενου ορισμού, το MRL, τότε εξορισμού πηγαίνει στο χαμηλότερο, στη χαμηλότερη εντοπίσιμη συγκέντρωση. Και το ερώτημα είναι ότι αν ακολουθήσουμε την προσέγγιση βάσει κινδύνου στις εξαιρέσεις, τι διαφορά θα υπάρχει. Και η απάντηση είναι που είναι ότι θεωρητικά θα μπορούσε, αλλά θα έπρεπε να αποδειχτεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από το MRL για την ανθρώπινη υγεία. Για μένα είναι πολύ δύσκολο να αποδειχτεί. Θα αξιολογηθεί με κάθε περίπτωση, χωριστά. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι από τις ουσίες που δεν έχουν ακόμα δοκιμιστεί βάσει αυτού αλλά θα κρεθούν ενδοκρινικοί διαταράκτες βάσει του ορισμού hazard base, δεν θα αυξηθεί το MRL, θα μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο και τελικά θα πρέπει να αξιολογούμε κατά περίπτωση Πάντως δεν υπάρχει καμία υπόνοια για το ότι θα αλλάξει το MRL και θα γίνει η τιμή του υψηλότερη. Το ζήτημα, τι άλλο ήταν, α, ναι, για τους ορισμούς είπαμε, για τον ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Δεν ε, μεταφράζεται κατά λέξη στο δικό μας κείμενο. Με αυτό που έχει σημασία είναι ο προτινόμενος ορισμός τι νόημα έχει, γιατί πρέπει να δουλέψουμε βάσει των ε, ορισμών που έχουμε τώρα για τα διοκτώνα κτλ. Συνεπώς εδώ έχουμε μία σωστή ερμηνεία του ορισμού της ΠΟΕ στο ευρωπαϊκό σύστημα. Τι άλλο. Πολύ υψηλά επίπεδα είπατε. Απόδειξης. Ίσως δεν ήμουν αρκετά ξεκάθαρος όταν σας εξήγησα τις αλλαγές που κάναμε στη διατύπωση. Γιατί αυτό το οποίο εξηγούσα σήμερα, οι αλλαγές στη διατύπωση, ήταν ακριβώς για να ανταποκριθούμε σε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι αλήθεια ότι ζητάμε δεν πρέπει να αποδεχτούν οι αρνητικέ συνέπειες επί του ανθρώπου. Πηγαίνουμε στα ίδια επίπεδα όπως έχουμε και με τον ορισμό της ΠΟΗ και βασιζόμαστε μόνο σε in vitro δοκιμές στα ζώα, αλλά επειδή το προηγούμενο σχέδιο είχε διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο όπου δεν φαινόταν από την πρώτη πρόταση, αλλά έπρεπε κανεί να διαβάσει δεν ξέρω πόσα άρθρα για να φτάσει εκεί. Τώρα το έχουμε κάνει πιο ξεκάθαρο το τι εννοούμε. Δεν ζητάμε δηλαδή αποδείξεις επί του ανθρώπου, δοκιμές δηλαδή επί του ανθρώπου, αλλά ότι αν η ουσία έχει δοκιμαστεί σε in vitro και στα ζώα και τα λοιπά, εντάξει. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Το επίπεδο δοκιμών είναι το ίδιο. Ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε συχνά εδώ είναι το θέμα της ε, ισχύω εν και το θέμα της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού μας τομέα. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ δύσκολη, ειλικρινά. Το βλέπετε και όλοι σας. Θα έπρεπε να είχαμε κάτι που να προστατεύει την ανθρώπινη υγεία χωρίς κανένα συμβιβασμό. Από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να σκοτώσουμε την ανταγωνιστικότητα του δικού μας αγροτικού τομέα απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν κάναμε την επιλογή να ακολουθήσουμε τον ορισμό hazard base και να μην συμπεριλάβουμε τον όρο potency, γιατί αυτό μας οδηγεί σε μια πολύ επικίνδυνη συζήτηση. Γιατί είναι ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο δρούν οι ουσίες αυτές και οι ενδοκρινικές ουσίες δρούν σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Μπορεί να πρόκειται για κάποια μόρια και είναι πολύ δύσκολο να πούμε που είναι το όριο. Συνεπώς, ο ορισμός είναι hazard base και γι' αυτό εμείς φτιάχνουμε αυτό το σύστημα και όχι το σύστημα potency. Η προσέγγιση βάση κινδύνου, risk δηλαδή, και όχι βάση βλάβης, hazard, είναι κάτι με το οποίο πειραματιζόμαστε σε πολλές άλλες ε, περιπτώσεις. Εδώ τώρα το δεχτήκαμε αυτό το επιχείρημα. Επίσης, αναρωτήθηκα εγώ ο ίδιος κατά πόσο συμφωνώ με αυτά που λέει η Εύσα. Ναι, είναι μια ερώτηση που είναι αξιόλογη, έχω τις απόψεις μου, αλλά υπενθυμίζω ότι οι συνομοθέτες πριν από χρόνια, αλλά και εσείς, αποφασίσατε ότι δεν είναι καλό αν είναι ο διαχειριστής κινδύνου που κάνει και την αξιολόγηση. Γι' αυτό και αποφασίσαμε την διαχείριση κινδύνου να τη χωρίσουμε από την εκτίμηση κινδύνου. Και αποφασίσαμε, το ένα θα γίνεται από την ΕΦΣΑ, ενώ η διαχείριση κινδύνου πρέπει να βασιστεί στην εκτίμηση κινδύνου. Συνεπώς, στη θέση που βρίσκομαι εγώ τώρα στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ δεν πρέπει να θέσω υπό αμφισβήτηση ή πώς να το πω, να κρίνω την επιστημονική αξία του σώματος το οποίο αξιολογεί. Εγώ, ό,τι μου λέει η ΕΦΣΑ, το θεωρώ επίσημη άποψη του δικού μας επιστημονικού σώματος και δουλεύω βάσει αυτής της πληροφορίας και μάλιστα πάμε ακόμα πιο μακριά και από αυτό γιατί πιστεύουμε ότι στη διαχείριση κινδύνου πρέπει να πηγαίνουμε πιο πέρα. Είπαμε ότι η διαχείριση κινδύνου είναι επαρκής, μάλλον δεν είναι αρκετή, και γι' αυτό πήγαμε και στην προσέγγιση βάση βλάβη ακριβώ εξαιτία τη συζήτηση που έχει γίνει για του ενδοκρινικού διαταράκτε. Συνεπώ, δεν θέλω να με βλέπετε σαν κάποιο που συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με την ΕΦΣΑ. Αυτό είναι ο ρόλο μου, να ακολουθώ τι δικέ του γνωμοδοτήσει. Και το τελευταίο που θέλω να πω και θα απαντήσει νομίζω και στις υπόλοιπες ερωτήσεις σας, είναι το εξή. Να υπενθυμίσω. Πολλές φορές υπόθηκε εδώ ότι φοβούμεθα ότι τελικά εν δυνάμει μπορεί να επιτρέψουμε να κυκλοφορήσουν ουσίες οι οποίες να είναι επικίνδυνες για καρκίνο ή για την αναπαραγωγή, για δεν ξέρω τι. Συνήθως αυτό λέμε για, τους, ε, για τις ουσίες τις ενδοκρινικές. Υπενθυμίζω όμως εδώ δύο πράγματα τα οποία τα γνωρίζετε έτσι κι αλλιώς πολύ καλά. Πρώτον, όλες οι ουσίες αξιολογούνται για τον κίνδυνο που ελοχεύουν πάντα, όλες. Και έτσι κι αλλιώς κανονικά καλύπτονται από εκεί. Μερικές φορές όμως είναι δύσκολη η αξιολόγηση και γι' αυτό η νομοθεσία έχει προβλέψει την υποχρέωση να κοιτάμε πιο συγκεκριμένα την, ε, το πόσο επικίνδυνε είναι οι ουσίες αυτές ε, για την αναπαραγωγή, για καρκίνο, για διάφορα. Οπότε, εδώ με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, αυτό που κάνουμε είναι ότι πολλαπλασιάζουμε την αρχή που έχουμε ήδη υιοθετήσει. Δηλαδή, μια ουσία που κινδυνεύει να είναι καρκινογενής δεν εγκρίνεται. Αυτό υπάρχει ήδη στην νομοθεσία μας. Όμως επειδή η ενδοκρινικός τρόπος δράσης μπορεί να τα ξεπερνάει όλα αυτά, έχουμε το σημερινό ορισμό. Αλλά δεν είναι αλήθεια ότι η τοξικότητα ή το κατά πόσο είναι καρκινογενής μειωσία ή όχι, είναι πράγματα τα οποία ε, δεν θα ισχύουν πια τόσο ισχύαν μέχρι τώρα εξαιτία του νέου ορισμού. Όχι. Ισχύουν αυτά τα κριτήρια έτσι κι και επεκτείνονται και σε άλλες δράσεις που ορίζονται ενδοκρινικά ενδεχομένως. Περί αυτού πρόκειται ο ορισμός. Και θυμάμαι πολύ καλά τη συζήτηση που γινόταν πριν τα αναλάβω εγώ αυτά τα θέματα. Είχε γίνει συζήτηση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και ποια ήταν η συζήτηση ότι αυτό που ήταν αρχικά ήταν. Θα ακολουθήσουμε τον ορισμό POI ή όχι, θα βασιστούμε στο hazard base ή όχι, αν ε, θα χρησιμοποιήσουμε το ενδυνάμει εφέ ή όχι. Σε όλα αυτά έχουμε πει ναι. Τα ακολουθούμε όλα αυτά που φαινόντουσαν να ήταν τα σωστά. Οπότε υπενθυμίζω πού βρισκόμασταν πριν από δύο χρόνια και πού βρισκόμαστε τώρα με την πρότασή μας ότι έχει καλύψει όλα αυτά. Ελπίζω λοιπόν, ελπίζω να απάντησα σε όλα τα σχόλια. Δεν θα σχολιάσω το ποιος πολιτικοποιεί τη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Well, thank you. Ευχαριστούμε πολύ, κύριο Μίκο. Σας ευχαριστώ γιατί πραγματικά αντιμετωπίσατε με πολύ θάρρος ε, το θέμα αυτό. Δεν είναι πάντα εύκολο τέτοια θέματα επίμαχα να συζητούνται σε αυτή την Επιτροπή. Θα παρακολουθήσουμε στενά το θέμα αυτό και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την πρόταση της Επιτροπής. Θα συνεχίσουμε όμως με το 15 σημείο της σημερινής διάταξης. Πρόκειται για τα λήματα ε, ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Αστικά Λύματα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με μια πολύ σύντομη παρουσίαση. Έχουμε και διαφάνειες. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ όποιος θέλει να βγει να το κάνει γρήγορα, λέει ο Πρόεδρος, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Με ησυχία. Thank you very much, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Λίγα λεπτά θα σας παρουσιάσω αυτά τα βασικά σημεία της έκθεσης. Ελπίζω να μπορέσω να, να αλλάξω και τη διαφάνεια. Να σας υπενθυμίσω καταρχήν τι είναι η οδηγία αυτή για τα αστικά αλήματα. Πριν από 20 χρόνια εγκρίθηκε και αρχικά ζητούμε από τις διάφορες αστικές περιοχές, κοινότητες, δήμους να συλλέξουν τα απόβλητα, να τα επεξεργαστούν και αυτό βάσει κάποιων συγκεκριμένων προδιαγραφών έτσι ώστε να αποφευθεί η ρήπανση ιδιαίτερα σε μεγάλες και πιο πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές και σε ευαίσθητες περιοχές. Κάτι δεν πάει καλά εδώ με το σύστημα για τις διαφάνειες. Θα ήθελα να γυρίσω στη διαφάνεια 2. Αυτοί που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα, υπάρχουν κάποια απορίσματα του ελεγκτικού συνεδρίου. Σας το λέω απλώς, αν θέλετε να κοιτάξετε με περισσότερη προσοχή πώς έχει εφαρμοστεί η οδηγία στις διαφορετικές χώρες όλα αυτά τα χρόνια, ποιες είναι οι απαραίτητες επενδύσεις. Βλέπετε εδώ αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε όλες αυτές τις ε, χρονικές ε, περίοδους που βλέπετε εδώ. Δεν μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε τα τελευταία στοιχεία για την Πολωνία. Η Κροατία επίσης δεν έχει συμπεριληφθεί, δεν ήταν υποχρεωμένη να μας στείλει τα τελευταία στοιχεία μετά την ένταξή της. Η επόμενη διαφάνεια. Δεν ξέρω αν βλέπετε εδώ την συλλογή λιμάτων. Λυπούμε, ίσως ε, δεν είναι σωστή ημερομηνία, εν πάση περιπτώσει, για τις 28 χώρες, για τις τελευταίες χώρες που προσχώρησαν υπήρχαν διαφορετικές υποχρεώσεις Γι' αυτό και υπάρχουν και δύο κατηγορίες όσον αφορά τις χώρες τις οποίες ισχύει αυτή η οδηγία περισσότερα χρόνια, για τις 15 δηλαδή, υπάρχει διαφορετική κατηγοριοποίηση συλλογής λιμάτων, διαφορετική επεξεργασία, αλλά λιγότερες υποχρεώσεις στις χώρες που προσχώρησαν αργότερα. Και αυτό εξηγεί βεβαίως η θέσει σε ισχύ αργότερα της οδηγίας εξηγεί αυτή τη διαφοροποίηση που βλέπετε. Αυτή είναι όμως η γενική εικόνα. Τι κάνει τώρα η Επιτροπή. Ουσιαστικά θα έλεγα κάνουμε τέσσερις διαφορετικές ε, δράσεις. Πρώτον, τη χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συναντούμε τα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε να λύσουμε θέματα διακυβέρνησης, διαχείρισης και ενδεχομένως υπάρχουν και οι προσφυγές, δικαστικές προσφυγές, περίπου 20 με διαφορα κρατημέλη. Εδώ θα ήθελα να σας δείξω στοιχεία που αφορούν, ε, αν θέλετε, τη γεωγραφική κατανομή της προηγούμενης ε, διαφάνειας. Είναι ίσως γραμμένα πολύ μικρά και δεν μπορείτε να διαβάσετε, αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι μπλε είναι καλό, με λίγα λόγια και τα κόκκινα είναι πολύ χαμηλή η συμμόρφωση και το κίτρινο είναι λίγο καλύτερο από το κόκκινο. Όπως σας είπα και προηγουμένως. Εδώ βλέπετε τις επενδύσεις. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί βεβαίως ε, είναι άμεσα συνδεδεμένες οι επενδύσεις και με την καλή υλοποίηση. Οι αριθμοί αυτοί βασίζονται σε εκτιμήσεις. 22 δις το χρόνο είναι το συνολικό ποσό που επενδύεται στον τομέα αυτό. 25% του ποσού αυτού χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια. 2015-2018 το ποσό αυτό θα αυξηθεί με 25 δισεκατομμύρια το χρόνο από 22 και βλέπουμε ότι υπάρχει μια σχετική βελτίωση των υποδομών που αφορούν τα αστικά λίματα. από τα από τη χρηματοδότηση ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Η χρηματοδότηση λοιπόν από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Ανοικοδόμηση Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνεισφέρουν στα έργα αυτά είναι για μας πάρα πολύ δύσκολο να μην έχουμε τα δεδομένα για να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί σε εσά αλλά και στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και βεβαίως σκοπός μας είναι να μειωθεί και το κόστος αυτών των επενδύσεων. Τέλος, κοιτούμε λίγο και την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρόκειται για νομοθεσία που αφορά το περιβάλλον, αλλά υπάρχει και πολύ σημαντικός οικονομικός αντίκτυπος. Πάνω από 600.000 θέσεις απασχόλησης. Ολοκληρώνω, νομίζω ότι μακρηγόρησα, αλλά είμαι και στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ λέει ο πρόεδρος. Ήταν πάρα πολύ σαφής η παρουσίασή σας. Θέλετε να πάρετε το λόγο, έχετε ερωτήσεις. Απευθύνομαι στους συναδέλφους της Επιτροπής. Ο κύριος Μπραντ. Θέλω κάτι να ρωτήσω που αφορά κάτι που συμβαίνει στις βόρειες χώρες και σίγουρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επειδή έχουμε την αλλαγή του κλίματος, έχουμε δυνατές βροχές σε σύντομες περιόδους. Περισσότερο από το παρελθόν και αυτό στο επιχειρηματικό σύστημα προκαλεί προβλήματα. Ακόμα χειρότερα έρχεται μετά το άλλο πρόβλημα. Έχουμε κάποιες περιοχές όπου θα ε, ρουφούσαν το νερό. Ας πούμε κάποιους ε, κήπους και κάποια πάρκιν. Όμως, κατά τη δεκαετία του 50 μέχρι τη δεκαετία του 70, ε, πήγε, μπήκε δάπεδο σε αυτές τις περιοχές. Έγιναν ε, πάρκινγκ τέλο πάντων. Βάλαν μπετόν. Και ενώ παλιά υπήρχε μόνο λίγο μπετόν για να πάει το αυτοκίνητο. Οπότε δεν είναι το νερό. Άρα βλέπουμε τώρα αυτή ο συνδυασμός του ότι δεν έχουμε απορροή των υδάτων, έχουμε περισσότερες βροχές και άρα και οι πορόδες περιοχές που τώρα έχουν έτσι δημιουργούν πρόβλημα. Έτσι γίνεται στο Εμένο Βασίλειο. Μήπως αυτό ισχύει και αλλού. We have also a request from Madame Dordano. Κύριε Ντορνάνο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσον αφορά την επεξεργασία αυτών των λιμάτων, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα με του υδάτινου πόρου και αυτό απειλεί τον πληθυσμό, ε, λένε και περισσότερο στι ε, αστικέ περιοχέ έχουμε 107 εκατομμύρια Ευρωπαίων που δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Επομένω, θα πρέπει να γίνεται καθαρισμό του νερού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό μια που είναι ένα πόρο σπάνια. Πάντω λέμε ότι οι περισσότερες ε, χώρες συμμορφώνονται προ την σχετική οδηγία για τα ελλείμματα και το σχετικό ε, κανονισμό παρά κάποια κενά που υπάρχουν όσον αφορά τη βιολογικό καθαρισμό. Οπότε λέμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με τους διαταράκτες, κάτι το οποίο είναι της καθής αλλά χρειάζεται ένα πρόγραμμα για τη συμμόρφωση, για τη χρησιμότητα. Μόνο έτσι είναι δυνατόν ε, ε, να προχωρήσουν οι τοπικές ε, αρχές, γιατί έχουν οικονομικά προβλήματα και γιατί δεν τους δίνει το κράτος χρήματα. Άρα χρειάζεται κάποιο θεσμικό, κανονιστικό πλαίσιο και για το τι γίνεται με τα δημόσια κτίρια. Ε, υπάρχουν εγγενισμοί, αλλά δεν μπορούν οι τοπικές ε, αρχές να, το, να, να ακολουθήσουν τα όσα επιτάσσονται. Άρα θα πρέπει αυτές οι νομοθετικές υποχρεώσεις να ξαλαφρώσουν για τις αρχές αυτές. Επίσης, για πετε μας τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την αξιολόγηση αξιούς των επιδόσεων των κρατών μελών τέλος πάντων. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν δεν έχει κανείς ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για το πρώτο ερώτημα. Ναι, είναι ένα πρόβλημα το ότι δεν υπάρχει απορροή των υδάτων όταν έχουμε καταγίδα. Είναι πρόβλημα αυτό σε όλες τις χώρες και μέχρι ενός βαθμού αυτό ρυθμίζεται, διότι δηλαδή υπάρχει υποχρέωση να διαχειριστεί κάποιο κράτος αυτό το πρόβλημα, όπως ξέρετε εσείς για τη δική σας χώρα. Υπήρχαν πάρα πολλές ένδικες ε, διαφορές και τελικά είχαμε εκτεταμένε επενδύσεις. Πάντως, με λίγα λόγια, όντως αυτό είναι πρόβλημα και το αντιμετωπίζουμε για να δούμε πώς θα βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη. Οι δύο και οι operators ήδη ο καθένας όσο μπορεί το αντιμετωπίζει. Και εμείς όσο μπορούμε από την πολιτική μας να προσπαθούμε να προωθήσουμε κάποια μέτρα. Και έχουμε και παραδείγματα όπου οι τοπικές αρχές και άλλοι εμπλεκόμενοι συνεργάζονται ώστε να εξασφαλίσουν το ότι υπάρχει λιγότερο τσιμέντομα και ούτως ώστε να μπορεί να υπάρξει απορροή των υδάτων. και να καταλήξουν το νερό αυτό στη θάλασσα. Να μην έχουμε επιπτώσει της μηνής στην υγεία, αλλά μην έχουμε πρόβλημα και για τις θάλασσες. Άρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αντιμετωπίζει το πρόβλημα, το εξετάζει, το αναγνωρίζουν τα κράτη-μέλη και μελετάτε του, τι μπορούμε να κάνουμε από πλευρά αναθεώρηση του νομοθετήματο. Τώρα για την άλλη ερώτηση. Είναι το θέμα σημαντικό. Δεύτερον, πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το τι μπορούν να κάνουν οι κοινοτικές δημοτικές αρχές, στην αρχή είχαμε βαθμία εφαρμογή της οδηγίας, γιατί ήταν μεγάλες υποχρεώσεις. Και έτσι αυξανόμενα, τέλος πάντων προοδευτικά, ε, επιβλήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές υποχρεώσεις και σε αυτές τις ε, τοπικές αρχές. Υποχρεώνται δηλαδή τα κρατημέλη να θεσπίσουν ισοδυνάμα μέτρα. Πάντως υπάρχει επικουρικότητα. Αλλά δεν μπορούμε να παρέμβουμε και να διατάξουμε το τι πρέπει να κάνουν οι αρχές. Πάντως υπάρχουν σοβαρές συνέπειες από το πρόβλημα, όπως τα είπατε. Ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας απαντήσατε και εδώ μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τελείωσε η συζήτηση για το θέμα. Το επόμενο είναι τα βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου. Είναι σχέδιο ψηφίσματος. Έχουμε εδώ τον κύριο Πότσα αλλά και τον κύριο Ντόφμαν όπως και την κυρία Ντορνανό. Οπότε μπορούμε να αρχίσουμε τη συζήτηση. You Ευχαριστώ πρόεδρε. και εγώ να ευχαριστήσω τους συναδελφούς για τις τρεις ψηφοφορίες ομόφωνα ενέκριναν τα κείμενα. Αυτό δεν το βλέπουμε καθημερινά στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πάνω όλους τους άλλους ε, συντάκτες των κειμένων. Όλες τι πολιτικές ομάδες υποστήριξαν τα ε, κείμενα μας. Οπότε τώρα μιλούμε για το ότι φαρμακευτικός κλάδος, όλοι οι μπλεκόμενοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να έχουμε μικρή έκθεση των τροφίμων σε βλαπτικές χημικές ουσίες. Οπότε θα πρέπει εδώ είπαμε να έχουμε κάποιο είδους ε, φυτοφάρμακα χαμηλού ρίσκου. Να δούμε τι θα γίνει με τα συνθετικά προϊόντα. Είπαμε όμως ότι από τις 7 ενεργές ουσίες οι 6 είναι βιολογικές θα πρέπει να δούμε το ότι επειδή θεωρούνται μικρή αποτελεσματικό, αποτελεσματικότητα και επειδή υπάρχει και γραφειοκρατία, δεν εγκρίνονται αυτές οι βιολογικές ουσίες. Όμως υπάρχει πρόβλημα εδώ για τους γεωργού, για όλο τον κόσμο και για το έδαφος ακόμα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ε, χρησιμοποιούμε αυτά τα βιολογικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου. Ο κανονισμός του 1107-2009 καλύπτει αυτές τις ουσίες, αλλά όχι όλες. Ούτε το ψήφισμα. Επίσης χρειάζεται κάποιο είδους προσαρμογή νομοθετική, ούτως ώστε να επιταχυνθεί η έγκριση αυτών των φυτοφαρμάκων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει λιγότερη γραφειοκρατία για τη διαδικασία έγκριση. Η προφορική ερώτηση βεβαίω και θέτει το ζήτημα νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων, ούτω ώστε να είναι πιο διαθέσιμα αυτά τα ε, φυτοφάρμακα. Όταν ήρθε των τροπολογιών, θα έχουμε πολλές γνώμες που θα προτείνετε, αλλά και η βιομηχανία θα ήθελε να δει ένα fitness check για το κατά πόσο δηλαδή σε δύο χρόνια ή να τον έχουμε αποτελέσματα η Κομισιόν όμως θέλει τη διαδικασία refit και να αντικατασταθεί εντελώς το 1107 Αυτό όμως χρειάζεται μία δεκαετία. Για μένα αυτό το fitness test θα πρέπει να άρει οποιασδήποτε αντιφάσεις ε, στους κανονισμούς. Ακριβώς αυτό ισχύει και για τον 1107 του 9. Γιατί δεν πέρα ε, δίνεται προτεραιότητα σε αυτά τα φυτόφαρμακα χαμηλού κινδύνου, αλλά δεν καλύπτονται κάποιοι μηχανισμοί ούτω ώστε να τους δίνεται προτεραιότητα στην πράξη. Γι' αυτό θέλω να μας πει πώς τα βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πρόεδρος. Χέρμπερτ, σε ευχαριστούμε. Η Επιτροπή. Όχι, ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Να ευχαριστήσω πραγματικά το συνάδελφο γιατί όπως είπε και ο συνάδελφος πως οι τροποποιήσεις του 2009 του αρχικού κειμένου πραγματικά ουσιαστικά για τα βιολογικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου και για όλες αυτές τις ουσίες υπάρχει μεγάλη υποστήριξη και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Φαίνεται εξάλλου και από την μέχρι τώρα πρόσκοπτη διαδικασία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επιτεχυνθεί και η διαδικασία για αυτά τα προϊόντα όσον αφορά την καταγραφή τους και την αδειοδότηση. Νομίζω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ταχεία αντίδραση και αυτό επιταχύνει και την παραγωγή και τη θέση στην αγορά. Όπως είπε και ο συνάδελφος θα πρέπει να περάσουμε στους απαραίτητους ελέγχους για να δούμε γιατί τον τελευταίο καιρό έχουμε δει πολλές προτάσεις από τον τομέα. Αυτός ο έλεγχος, fitness check, να βελτιώσει την νομοθεσία, κάτι που νομίζω όλοι το υποστηρίζουν και θα πρέπει να δούμε με μεγάλη προσοχή αν αυτή η διαδικασία επιτάχυνσης είναι κάτι που μπορούμε να το πετύχουμε ή όχι. Βεβαίως ε, εδώ δεν αναφερόμαστε σε μεγάλες επιχειρήσεις, ε, πρόκειται για μικρομεσαίες ε, εταιρείες και πολλές φορές τους λείπουν τα χρήματα για να μπορέσουν να στηρίξουν αυτές τις ταχείες διαδικασίες εγγραφής και διάθεσης στην αγορά. Νομίζω θα πρέπει να τους προσφέρουμε εναλλακτικές ε, διαδικασίες έτσι ώστε αυτά τα βιολογικά φυτοφάρμακα, τα εναλλακτικά να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από τους καταναλωτές. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το πολύ θετικό και για την υγεία και από τη στιγμή που είδαμε αυτή την πολύ θετική ψηφοφορία σήμερα το πρωί νομίζω ότι μπορεί να είμαστε αισιόδοξη και να βρεθεί μια γρήγορη λύση, όπως είπε ο συνάδελφος Πώς. Έχει κρατήσει πολλά χρόνια αυτή η διαδικασία και δεν έχουμε στηρίξει ε, το τομέα. Ήρθε η ώρα νομίζω να δράσουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντόρνανό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σαν συνεισηγήτρια του κειμένου αυτού θα ήθελα και εγώ να διευκρινίσω κάτι, ιδιαίτερα όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία, όσον αφορά τα παραδοσιακά φυτοφάρμακα. Από τη μία έχουμε τους αγρότες, τους γεωργούς και από την άλλη τους υπόλοιπους καταναλωτές και Ευρωπαίους πολίτες. Αυτοί που απειλούνται κυρίω είναι η πρώτη κατηγορία, οι αγρότε και οι γεωργοί που είναι σε άμεση επαφή με αυτά τα χημικά φυτοφάρμακα. Όσον αφορά τώρα την ε, χημική αυτή, ε, τις χημικές αυτές ουσίες και τη χρήση τους στην βιολογική γεωργία και την ε, άρση των απαγορεύσεων, είναι κάτι που θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να το συζητήσουμε. Πρέπει να προστατεύσουμε τον τομέα της βιολογικής παραγωγής και καλλιέργειας, καθώς και την υγεία των γεωργών και των καταναλωτών μας. Πριν την θέση στην αγορά και την ε, εμπορική διάθεση αυτών των φυτοφαρμάκων, θα πρέπει η εγγραφή τους, η καταγραφή τους και η αδειοδότησή τους να γίνει με εξαιρετική προσοχή επικρατεί ένα ολιγοπόλιο στον τομέα αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εισχωρήσουν ανταγωνιστές, ιδιαίτερα κάποιοι νέο εισαγόμενοι οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν βιολογικά φυτοφάρμακα. Είναι μεγάλη η πίεση των μεγάλων επιχειρήσεων. Κοιτάξτε παραδείγματος χάρη την Bayer που συγχωνεύθηκε πολύ πρόσφατα με την Monsanto η χρήση των βιολογικών φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου δεν είναι κάτι που το ζητούν τα κράτη-μέλη. Η πραγματική αιτία είναι ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ανάπτυξη αυτού του τομέα σήμερα, αυτά τα βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου είναι λιγότερο αποτελεσματικά λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης και στήριξής τους από απαραίτητες δομές και μέσα. Θα πρέπει τα βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου να τα στηρίξουμε. Ήρθε η ώρα να δράσουμε. Δεν νομίζω πλέον ότι έχουμε χρόνο να συζητήσουμε για την ανάγκη να στηρίξουμε τα βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου και την διάθεσή τους στην αγορά. Ίσως θα ήταν σωστό να υπενθυμίσω ότι μία ομάδα εκπροσώπων της ΕΦΣΑ και των κρατών μελών έχουν βεβαίω συμμετάσχει στη διαδικασία πρόθεση και στήριξη των βιολογικών φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου. Θα υπενθυμίσω και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών που είναι η παραγωγή φυτοφαρμάκων με αυτές τις δραστικές ουσίες. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπονομεύσουμε εδώ και να υποτιμήσουμε τις δυνατότητες και αρμοδιότητες των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Ευχαριστούμε. Άλλοι ομιλητές? Όχι. Ο κύριος, ο ε, ε, κυρία Λάι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να επιστήσω την ε, προσοχή σας, λέει κυρία Ντελέ, στο ότι υπάρχουν πολλές αντιθέσεις, φυτογενομικά προϊόντα, ε, χημικά και φιολογικά έχουν ε, μεγάλη διαφορά. Η συζήτηση αυτή λοιπόν μας θυμίζει μια δογματική συζήτηση και όχι ρεαλιστική. Στο κάτω-κάτω η φύση έχει δημιουργήσει τις περισσότερες ουσίες και όχι η πετροχημική βιομηχανία. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί και για τα προϊόντα αυτά, τα βιολογικά χαμηλού κινδύνου, να τους κρατήσουμε τη θέση που τους πρέπει. Είναι κίνδυνο να τα παράγουμε και να τα επιτρέπουμε χωρίς χρονικό όριο. Πρέπει κάθε τόσο να ελέγχουμε και πάλι. Να ενθαρρύνουμε επίσης την έρευνα και την αδειοδότηση για την διάθεση στην αγορά πρέπει να γίνεται κάθε τόσο, τόσο για τα βιολογικά όσο και για τα κλασικά. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε βεβαίως και καινοτομίε για τα παρασιτοκτόνα, χωρίς να επιβάλλουμε ημέν τις λύσεις μας στους δε, δεδομένου μάλιστα ότι οι αγρότες σήμερα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέψουν τι θα τους συμβεί στο μέλλον. Ενθαρρύνω λοιπόν τις χώρες μέλη να ανταλλάξουν πληροφορίες επί του θέματος όσο γίνεται περισσότερο μεταξύ του. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ο κύριος Μπάτσο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ζήτησα τώρα το λόγο γιατί τώρα μου ήρθε μια ερώτηση. Πολύ σύντομα. Θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας από τα αέρια του θερμοκηπίου. Και πιστεύουμε ότι είναι αυτό τόσο σημαντικό που είμαστε διατεθειμένοι να επιδοτήσουμε τεχνολογίες οι οποίες δεν απελευθερώνουν άνθρακα, ολική ενέργεια, ηλιακή κτλ. Αλλά από αυτό ακολουθεί η εξή ερώτηση. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη υγεία, έτσι δεν είναι. Άρα πρέπει να προωθήσουμε βιολογικά παρασιτοκτόνα. Υπάρχει κάτι που να μας εμποδίσει να επιδοτήσουμε τη χρήση τέτοιων παρασιτοκτόνων βιολογικών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Υπάρχει άλλη ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα παρασιτοκτόνα αυτά, τα βιολογικά χαμηλού κινδύνου. Όχι. Ωραία. Thank you, Chair. Ladies and gentlemen, the Commission welcomes this this discussion and also the content of the. Η Επιτροπή χαίρεται για τη συζήτηση αυτή. Ακούστηκαν διάφορες ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές. σχόλια, παρατηρήσεις. Πολλά από αυτά έχουν ληφθεί υπόψη. για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας υπενθυμίσω την ίδια την αρχή της νομοθεσίας. Η έγκριση ουσιών που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνα, είτε πρόκειται για συνθετικές ουσίες είτε για βιολογικές, γίνεται άπαξ και ουσίε αυτές έχουν περάσει από αξιολόγηση κινδύνου. Εδώ δεν κάνουμε διάκριση. Το σύστημα δεν κάνει διάκριση της αξιολόγησης κινδύνου για τα βιολογικά και τα συνθετικά προϊόντα, τις ουσίες. Είναι ίδια η αξιολόγηση. Παίρνει χρόνο, κοστίζει Η αξιολόγηση λοιπόν δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στα βιολογικά και τα συνθετικά παρασιτοκτόνα. Έχουμε όμως διαφορετικές απαιτήσει για τα δύο είδη αυτά ουσιών. Μετά από την επιτυχή αξιολόγηση μπορεί να ταξινομηθεί ως χαμηλού κινδύνου ένα φυτοφάρμακο. Προβλέπονται λοιπόν χαμηλού κινδύνου, αλλά υπάρχει και μια κατηγορία που ονομάζεται βασικές ουσίες και μετά υπάρχει μια μεγάλη ομάδα συνθετικών μυαλών. Η ταξινόμηση αυτή χαμηλού κινδύνου ουσίες δεν κάνει διάκριση, όπως είπα, ανάμεσα στα βιολογικά και τα συνθετικά παρασιτοκτόνα. Το τρέχον σύστημα, έτσι όπως έχει στην νομοθεσία μας σήμερα, επιτρέπει και στις συνθετικές ουσίες, όπως και στις βιολογικές ουσίες, να μπορούν να κριθούν ότι είναι χαμηλού κινδύνου ουσίες. Βέβαια, η ορολογία μιλάει για βιολογικά χαμηλού κινδύνου. Για μας δεν υπάρχει αυτό. Όπως επίσης και η βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων παριστοκτόνων. Εδώ το κείμενο χρησιμοποιεί μόνο τον όρο χαμηλού κινδύνου ουσίες. Το κείμενο, το σχέδιο αναφέρει διάφορες περιπτώσεις και απευθύνεται σε οργανώσεις, χώρες και τα λοιπά για να επιταχυθεί η διαδικασία και ώστε οι ουσίες χαμηλού κινδύνου, βιολογικές, να τεθούν γρήγορα στην αγορά. Κάποιες από αυτές έχουν μπει ήδη στη διαδικασία. Με την Ολλανδική Προεδρία ήδη συζητήσαμε κάποιες από τις πτυχές και συμφωνήσαμε ότι με την τρέχουσα Προεδρία θα έχουμε ένα σχέδιο για να προωθήσουμε βιώσιμες ουσίες. Όλα αυτά μέσα στα πλαίσια του σημερινού νομικού πλαισίου Έχουμε αναθεωρήσει τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των ουσιών ως χαμηλού κινδύνου. Είχαν εγκριθεί καταρχήν το 2009 και διορθώθηκαν για να καλύψουν και βιολογικές ουσίες ως χαμηλού κινδύνου. Αναθεωρούνται λοιπόν τα κριτήρια, υπάρχει ένα σχέδιο ήδη που διευκρινίζει διάφορες πτυχές. Μιλάει για μικροοργανισμούς που έτσι καλώς μπορούν να θεωρηθούν εξορισμού χαμηλού κινδύνου. Υπάρχει ένας μηχανισμός feedback, ανάδρασης, Δηλαδή γίνεται διαβούλευση με τον κόσμο, γίνεται ψηφοφορία. Έτσι κι αλλιώς έχουμε συνεργαστεί με πολλούς φορείς, όχι μόνο από τον χώρο της Γεωργίας, αλλά με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και το κοινό γενικά, για να εγκριθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτή η τροποποίηση και θα ελεγχθεί βεβαίω από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μια άλλη δραστηριότητα για να προωθήσουμε τα, τις ουσίες χαμηλού κινδύνου είναι ότι πολλές ουσίες μπορούν εν δυνάμει να θεωρηθούν χαμηλού κινδύνου που εγκρίθηκαν πριν από 10 χρόνια όταν δεν υπήρχαν ίδιες κατηγορίες και δεν υπήρχε το ίδιο επίπεδο ταξινόμησης. Υπάρχουν ήδη πολλά φυτοφάρμακα στην αγορά και τα προϊόντα αυτά, οι ουσίες, έχουν μια περίοδο έγκρισης δεκαετή. Μετά υπάρχει ανανέωση και στην ανανέωση αυτή θα δώσουμε προτεραιότητα στις ουσίες εκείνες όπου η Επιτροπή με εμπειρογνώμονες είπαν ότι είναι δυνάμει ουσίες χαμηλού κινδύνου. Οπότε θα υποφεληθούμε πιο γρήγορα μέσω της νομοθετικής διαδικασίας. Και για να καλύψουμε το διάστημα από τώρα μέχρι την ανανέωση των ουσιών αυτών. Όπως σας είπα, η διαδικασία είναι πάρα πολύ περίπλοκη και παίρνει χρόνο, είναι χρονοβόρα. Για να καλυφθεί πάντως αυτό το χρονικό διάστημα, σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε ένα μη δεσμευτικό κατάλογο δυνάμει χαμηλού κινδύνου ουσιών, που θα επιτρέψουν στις χώρες μέλη, αν μη τι άλλο, να δουν τις δικές τους διαδικασίες αξιολόγησης σε θελοντική βάση και να χρησιμοποιήσουν τις ουσίες ε, αυτές. Κάτι άλλο. Αναφερθήκατε στο πρόβλημα της αποτελεσματικότητας των ουσιών αυτών, που συνήθως είναι χαμηλότερη από ό,τι εκείνη των χημικών φυτοφαρμάκων. Η οργάνωση προστασίας που δεν περιλαμβάνει μόνο χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλες ανατολικές χώρες ή της Μεσογείου ετοιμάζει νέες κατευθυντήριες γραμμές για να επιτρέψει μια καλύτερη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου. Κάτι που περιμένουμε να έχουμε μέχρι τα τέλη της επόμενης χρονιάς. Ρωτήσατε για το REFIT. Η Επιτροπή αποφάσισε όλη την νομοθεσία για τα φυτοφάρμακα να την υποβάλει στο REFIT. Δεν αποφασίσαμε για fitness check, Για το Refit, ο χάρτης πορείας λέει ότι γίνεται δημόσια διαβούλευση και περιμένουμε σχόλια για να προχωρήσουμε σε έγκριση. Επίσης, εκφράστηκε επιθυμία να υπάρξει ορισμός για τα βιολογικά χαμηλού κινδύνου. Θα γίνει στο μέλλον, σε μελλοντική νομοθεσία. Προς το παρόν δεν έχουμε νομοθετικές ρυθμίσεις για αυτή την κατηγορία προστασίας. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα και ελπίζουμε να έχουμε αποτελέσματα μέσα στο πρώτο εξάμενο του 2017. Η βασική αρχή παραμένει ότι η ουσία πρέπει να αξιολογηθεί ως προς την επικίνδυνοτητά της να περάσει αυτές τις εξετάσεις επιτυχώς και όσον αφορά τα ζώα και όσον αφορά τον άνθρωπο. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε που απαντήσατε στις ερωτήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα κάνουμε διακοπή στη συνεδρίασή μας. Διακοπή μέχρι τις 5.30. Γιατί τότε θα συζητήσουν το τελευταίο σημείο της μεσδιαταξιός, δηλαδή ανταλλαγή απόψεων τον κύριο Ντανιέλ Καγέχα Κράσπο για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Επομένως, Διακόπτουμε μέχρι τις 5.30. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Dear colleagues, dear General Director. Αγαπητοί συνάδελφοι, Γενική Διευθυντά, περιμέναμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να αρχίσουμε. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Διευθυντή Τανιέλ Καγέχα Κρέσπο όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Νοεμβρίου ενέκρινε ένα πακέτο για την εφαρμογή των στόχων ε, για την ανάπτυξη. Υπάρχει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά είναι καλύτερα να τα ακούμε απευθείας από τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος. Τι αποφασίσαμε λοιπόν Σήμερα το πρωί οι συντονιστές αποφάσισαν να αρχίσουν μια έκθεση πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό. Και πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε στο μέλλον. Πάντως τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ακούσουμε την παρουσίασή σας και μετά φυσικά θα αντιδράσουμε κι εμείς. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ε, παρουσίασή σας και με μεγάλη μου χαρά να σας παρουσιάσω τις αδρές γραμμές αυτής της ανακοίνωσης της Επιτροπής για τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Επιτρέψτε μου να αρχίσω υπενθυμίζοντας όπως γνωρίζετε αυτή την ε, έγκριση από τον ΟΗΕ τη θεματολόγη του 2030 για αυτούς τους στόχους. Το Σεπτέμβριο του 10 αυτό ήταν ε, ένα ορόσημο, ήταν ένα επίτευγμα, διότι για πρώτη φορά έχουμε μια τέτοια συνολική οπτική όσον αφορά τη βιώσιμη ανέβριση για όλους. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ε, αυτό ε, συνεκέντρωσε το ναι όλων των ε, κρατών μελών του ΟΗΕ. Και επίσης λέω ότι είναι ορόσημο και για ένα άλλο λόγο, γιατί έγινε διαπραγμάτευση με όλους τους εμπλεκομένους. Με αυτό το θεματολόγιο έγινε μια στροφή. Στροφή από τους στόχους της ε, χιλιετίας που είχαμε τις πιο ανεπτυγμένες χώρες που συνεργάστηκαν με τις ε, αναπτυσσόμενες. Τώρα όμως έχουμε... Ε, ναι. Έχουμε αυτούς τους 17 στόχους 169 σχετιζόμενους ε, υποστόχους και καλύπτουμε πολιτικές από την ε, παινία μέχρι την διατροφική ασφάλεια, μέχρι την βιώσιμη ανάπτυξη και θέματα περιβάλλοντος. Το νερό, την ε, χωροταξική ανάπτυξη των πόλεων, την θάλασσα και αποτελεσματική χρήση των πόρων. Δεν ε, πρόκειτο για ένα ακόμα ψήφισμα. πρόκειται πρόκειτο για πολιτική δέσμευση που θα οδηγήσει σε ανάληψη δράσης. Δεν ήταν ακόμα μία διακήρυξη δήλωση, ήταν μία κοινά ε, αναληφθήσα υποχρέωση σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε τοπικό και σε ευρωπαϊκό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο σε σχέση με αυτή την συναυτήσα συμφωνία. Γιατί? Διότι έχει δεσμευτεί για την βιώσιμη ανάπτυξη. Την έχουμε εντάξει στις προτεραιότητες και στις πολιτικές μας. Και επίση, με περηφάνεια θεωρήσαμε ότι είμαστε πρωτοπόροι για να συναρθεί αυτή η συμφωνία και σας τονίζω ότι αυτό που θέλουμε είναι να συνεχίσουμε να είμαστε πρωτοπόροι όσον αφορά την βιωσιμότητα. Και για αυτό, σε αυτή τη φάση και τη μόλις περασμένη εβδομάδα εγκρίναμε αυτό το οποίο αναφέρατε, Πρόεδρε. Τη δέσμη μέτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τρεις ανακοινώσεις. Πρώτα-πρώτα για τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, Δεύτερον, την Ευρωπαϊκή Συνένεση για Ανάπτυξη, που αποτελεί ένα προσχέδιο πολιτικής για ανάπτυξη. Και το θεματολόγιο, το οποίο έπεται του τέλους της ε, κότονου σχέσης δηλαδή με Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικό. Οπότε και προχωρώ στα της ανακοίνωσης για την ανάπτυξη, γιατί παρά το ότι όλοι αυτοί οι δεσμοί μέτρων είναι μια σφαιρική ε, ανταπόκριση και θεώρηση κομισιών ότι είναι σωστό να έχουμε εξωτερική διάσταση και εξωτερική διάσταση όμως ο, παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καλύψουμε τα επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη. Γι' αυτό και αυτό το ονομάσαμε το ευρύτερο πλαίσιο της στέγη αυτών των ε, ε, νομοθετημάτων και προτεραιοτήτων για την Επιτροπή. Οπότε επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι αφετηρία αποτελεί το ότι η Ευρώπη δεν είναι σε κακή θέση για να πετύχει τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης γιατί οι πολιτικές μας σήμερα ε, αποσκοπούν και ευθυγραμμίζονται με αυτούς τους στόχους. Άρα μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι. Το Δευρωματικό Κοινοβούλιο μπορεί να αξιώσει μια μερίδα ε, αυτού του πιτεύματος γιατί χάρη στο έργο το οποίο επιτελείται η Ευρώπη βρίσκεται σε καλύτερη θέση από όσο θα ήταν αν απουσίσουν αυτά τα στοιχεία όμως αυτά όλα είναι επιτεύγματα αυτά όλα είναι πρόοδος αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ότι έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή και η στοχευμένη δράση σε όλους τους τομείς. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε παρά το ότι είμαστε πιο μπροστά από άλλε περιοχέ του κόσμου, τότε θα έχουμε πρόβλημα, δεν θα πετύχουμε τους στόχους. Η Επιτροπή στην ανακοίνωση αυτή ε, αναφέρει ποια είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί στο εγγύς Μετά από σκληρή δουλειά, επικεφαλής ήταν ο αντιπρόεδρος Τίμερ και έχουμε και ένα project team 20 επιτρόπων για την ε, πολιτική καθοδήγηση και σα ενημερώνω ότι ο Τίμερμαντς θα συνεχίσει με την ίδια ομάδα και έτσι να υπάρχει πολιτική συνέχεια για όλους τους τομείς. Τώρα ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το ότι θα πρέπει να χαράσετε πολιτική επί τη βάση δείξεων, αποδείξεων, στοιχείων και για να ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα θα πρέπει να είμαι θα εστέσεν, να κάνουμε προσαρμογές, να ε, ε, είμαστε υπόλογοι σε κοινοβούλιο, σε Ευρωπαίους και ε, να μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε έκθεση πρόοδου πεπραγμένων και σε σχέση με όλους τους εταίρους μας επίσης να μπορούμε να αναφερόμεθα και στον ε, ΟΗΕ. Και όσον αφορά τώρα το περιβάλλον, έχουμε μία ανακοίνωση που δίνει μεγάλη σημασία σε αυτή τη διάσταση και ευθύ εξ αρχή αναφέρεται. Η οπτική της ε, Ευρώπης σημαίνει αξιοπρέπεια για όλους, σε όλο τον πλανήτη. Αλλά θα πρέπει να συγκεράσουμε ευημερία, αποτελεσματικότητα, η ελληνική κοινωνία, να μην περιθωριοποιείται κανένας και υπεύθυνη θέση για το περιβάλλον. Η υλοποίηση του κεκτημένου θα οδηγήσει στην βιωσιμότητα. Θα πρέπει βέβαια να επαναλάβουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι περίπλοκη, γιατί έχουμε πάρα πολλούς στόχους, πάρα πολλές πολιτικές που σχετίζονται με αυτούς. Οπότε με αυτή την ανακοίνωση προσπαθούμε να κάνουμε μια καταγραφή αυτών των πολιτικών, να διαπιστώσουμε το πού βρισκόμαστε σε σχέση με την επιτευχή των στόχων. Και αυτή η καταγραφή έριξε ότι βέβαια υπάρχουν κανονισμοί που καλύπτουν αυτή την πορεία σε σχέση με τους φυσικούς πόρους. Αλλά επίσης έτσι καταλάβαμε ότι αναγνωρίζεται το πόσο σημαντική είναι η προστασία των εθνικών πόρων για να πετύχουμε τους στόχους μας. Οπότε Σαν παράδειγμα να αναφέρουμε το πόσο σημαντική είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Θα πρέπει αυτή να εστιάζεται όλο ένα περισσότερο στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων σε σχέση και με το κλίμα. Έτσι θα πετύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Και παρομοίως η ελευτική πολιτική θα πρέπει να βοηθά στη βιωσιμότητα της ε, αλίας. Οι πολιτικές υγείας να λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά με το περιβάλλον, αλλά και η κυκλική οικονομία. Αποσυνδέει την οικονομική ανάπτυξη από την καταστροφή του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζεται ως ε, απειλή, και κοινό στοιχείο σε όλα τα θέματα, είναι η βιωσιμότητα σε σχέση με την ε, ένταξή της σε όλες τις πολιτικές. Να το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Και αυτό που θέλει να στείλει ο κύριος Τίμερμανς, βιωσιμότητα, θα πρέπει να σημαίνει ο μπούσουλος για ε, όλο μας το έργο. Εάν θέλουμε το μέλλον για τον πλανήτη και για τα παιδιά μας να είναι αυτό που χρειάζεται. Σε σχέση επίσης και με το θεμελό του 2030. Πρόκειται για δέσμευση όλων και άρα όλοι πρέπει να βοηθήσουν. Επίσης στην ανακοίνωση αναγνωρίζεται ότι δεν χρειάζεται δράση μόνο από πλευρά κομισιών. Πρέπει να συνεργαστούμε το Κοινοβούλιο με όλα τα θεσμικά όργανα. Αλλά και τα κρατημέλη φέρουν ευθύνη για τους τομείς αρμοδιότητας. Επίσης αναγνωρίζεται η συμβολή του ιδιωτικού τομέα του επιχειρηματικού κόσμου για αυτούς τους στόχους υπέρ του περιβάλλοντος. Και άρα χρειάζεται ανάλογη συμπεριφορά των επιχειρήσεων για όλες τις προκλήσεις της κοινωνία και του περιβάλλοντος. Κάτι άλλο επίσης πάρα πολύ σημαντικό που μπορεί και μας απασχολεί περισσότερο στον ΟΗΕ έχουμε μια έκθεση. Τι γίνεται με το χρηματοπιστικό σύστημα, πώς θα πρασινίζει. Green Finance. Πρέπει να είναι και βιώσιμα τα χρηματοοικονομικά. Άρα αυτό έρχεται να σχετιστεί με τους στόχους. Οπότε και εμείς τονίσαμε το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει σχετικό ψήφισμα. Άρα ε, ακολουθούμε το μήκο κύματο το δικό σα. Τώρα, θα πρέπει να γίνουν ε, έργα, θα πρέπει να αναπτυχθεί προ δύο κατευθύνσει. Για το θεματολόγιο του 2030 θα πρέπει αυτοί οι στόχοι να ενταχθούν στο θεματολόγιο και του 2020. Το συζητήσαμε αυτό και έχουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, έχουμε το θεματολόγιο 2020, έχουμε το 7ο ε, περιβαλλοντικό πρόγραμμα, έχουμε τώρα τους στόχους του 2030, αλλά όλα αυτά θα πρέπει μεταξύ τους να έχουν κάποια συνοχή και συνέπεια. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Πρώτα-πρώτα ανταπόκριση άμεση και να εγκρίνουμε αυτούς τους στόχους τους βιώσιμους ε, στο θεματολόγιο του 2020. Επίσης θα πρέπει να ξεκινήσουμε ανάληψη δράσης μακρόπνοα, δηλαδή και μετά το 2020. Επομένως, θα πρέπει ε, όλες αυτές οι επιμέρους κατευθύνσεις να συγκεραστούν. Οπότε να, και τώρα αναδύεται η σημασία του νέου πολιτισμού μεσού πλαισίου μετά το 2020. Γιατί θα πρέπει να δοθεί κατεύθυνση τέτοια που να εξασφαλίζει ότι ο κοινοτικό προπολογισμό και αυτό βοηθάει στην επίτευξη αυτών των μακρόπνων στόχων. Υλοποίηση τώρα του θεματολογίου του 2030. Αυτό είναι κοινή ευθύνη. Άρα σας τονίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή να έχει υπόψη της τις απόψεις σας, προτάσεις βελτίωσης αυτής της υλοποίησης και οπωσδήποτε θα πρέπει το Κοινοβούλιο να βοηθήσει σε αυτή την υλοποίηση. Άρα θα πρέπει να υπάρξει συνειδητοποίηση της ανάγκης ε, της βιωσιμότητας ε, αυτό να φτάσει στα κράτη-μέλη. Είπαμε θα εμπλακούν όλοι οι επίτροποι και επίσης να εμπλακούν όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και ξέρω ότι σε αυτό συμφωνείτε και θα το κάνετε. Επίσης λέμε ότι πρόκειται για κοινό θεματολόγιο. Αφορούν τους ε, Ευρωπαίους, την κοινωνία των πολιτών, τις οργανώσεις, ε, τις επιχειρήσεις. Όλοι δεν έχουν ρόλο να παίξουν, όλων η φωνή πρέπει να ακουστεί και έτσι να έχουμε μια πλατφόρμα που να συγκροτήσουμε και να υπάρξει προετοιμασία θα έχουμε στις 20 Δεκεμβρίου μια συνάντηση υψηλού επίπεδου με στόχο τη δημιουργία αυτής της πλατφόρμας. Νομίζω ότι πέραν να σας λέω, θα ακούσω και τις ερωτήσεις σας, γιατί την ανακοίνωση την έχετε διαβάσει. Η ανακοίνωση, θέλω να σας πω ότι είναι απλώς μια αφετηρία. Μην περιμένετε ότι εκεί μέσα δίνουμε απαντήσεις σε όλα τα θέματα. Αλλά το, το οποίο μετράει είναι τι δράση θα αναλυθεί στη συνέχεια. Υπάρχουν εδώ έξι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία όσον αφορά την διαδικασία και την πορεία. Εμείς πρόκειται να εντάξουμε αυτούς τους στόχους σε όλες τις μεσοπρόθεσμες πολιτικές. Αυτό θα πρέπει να γίνει για πάσα υπάρχουσα πολιτική. Για να έχουμε υπόψη ομένως τους, τους τρεις ε, γιώνες, τους τρεις πυλώνες. Ε, οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον. Επίσης, από το 2020 και μετά πρόκειται να έχουμε τακτές εκθέσεις για το πώς υλοποιούνται αυτοί οι στόχοι. Είναι σημαντικό να υπάρξει παρακολούθηση, να δούμε αν υπάρχει πρόοδος ή ου. Κατά τρίτο λόγο θα συνεχίσουμε να συνοούμαστε με τους εξωτερικούς εταίρους γιατί οι βιώσιμοι στόχοι δεν είναι θέμα μόνο ευρωπαϊκό. Θα πρέπει να υπάρξει αναπτυξιακή συνεργασία με τον υπόλοιπο κόσμο. Κατά τέταρτον θα θέλαμε να υλοποιήσουμε το θεματολόγιο 2030 σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Να, ως παράδειγμα σας αναφέρω ότι η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση είναι σημαντικός στόχος. Να, που ωφελεί η κυκλική οικονομία και να που χρειάζεται η σύμπραξη του Κοινοβουλίου. Οπότε θα πρέπει να έχουμε αυτή την πλατφόρμα ε, όλων των εμπλεκομένων που σας ανέφερα και έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε ανταλλαγή των καλύτερων ε, πρακτικών για την υλοποίηση σε όλους τους τομείς. Και τελευταίο και σημαντικό κινούμεθα παράλληλα για την περίοδο ως προοπτική μετά το 2020 και γνωρίζουμε ότι πρόκειται μόνο για μια πρώτη φάση και ότι και άλλα θα ακολουθήσουν. Όμως θεωρούμε ότι με αυτή τη δέσμη μέτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρόκειται να μπει σε νέο δρόμο η, κίνησή μας μέσα στην παγκόσμια οικονομία και είναι κάτι αυτό για το οποίο όλοι έχουμε δεσμευτεί. Γι' αυτό και εγώ θέλω να ακούσω τις απόψεις τις δικές σας και γνωρίζουμε ότι το Κοινοβούλιο συμμερίζεται τις ε, φιλοδοξίες μας για το θέμα του 2030 και η βιωσιμότητα ε, γεννήθηκε εδώ στην Ευρώπη και σας βεβαιώ ότι εκτιμώ πάρα πολύ τις προτάσεις σας και τη δουλειά σας άρα να πώς θα βελτιώσουμε τη διαδικασία αυτή ως τη γνώμη σας ε, κάτι θα λείπει είπαμε είναι υψηλές οι φιλοδοξίες αλλά μπορείτε να τα βελτιώσετε όλα. Να δούμε πώς θα συνεργαστούμε με τα θεσμικά όργανα. Όλα αυτά είναι ζητήματα. Εμείς απλώς θέλουμε να δώσουμε το ανακτήριο λάκτισμα για μια συζήτηση και με τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια διαδρομή στην οποία όλοι θα συμμετάσχουν. Και στο τέλος θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, τόσο σημαντική πρόκληση. Την υλοποίηση του θεματολογίου 2030, κάτι το οποίο είναι το κλειδί για το μέλλον των ε, Ευρωπαίων. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now we can uh, start. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιούζο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον Γενικό Διευθυντή που ήρθε να μας εξηγήσει σήμερα τις ανακοινώσεις αυτές. Δίνω συγχαρητήρια στην Επιτροπή που είναι φιλόδοξη, που έχει αυτούς τους στόχους που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικοί. Η Ευρώπη μπορεί να τους πετύχει. Έχει σαν βάση τις προτάσεις για την κυκλική οικονομία, για τη μείωση των εκπομπών εκεί που δεν υπάρχει το θέμα των πληστηριασμών δικαιωμάτων. Είμαι σίγουρη λοιπόν ότι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος εδώ θα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον καλύτερο σύμμαχο. Καλωσορίζω και την πλατφόρμα που μας παρουσίασε. Όντως πρέπει να δοθεί συνέχεια σε όλους αυτούς τους στόχους. Πώς εντάσσεται η επιχειρηματική κοινότητα, ρωτάτε. Νομίζω ότι αν δει τα ωφέλη για την οικονομική της ανάπτυξη, η κοινότητα αυτή θα ενταχθεί αμέσως. Και θα το δει αν υπάρξουν μέτρα τα οποία βελτιώνουν το περιβάλλον, θα βελτιώνεται και η τεχνολογία, οπότε αυτό θα είναι κέρδος και για τις επιχειρήσεις. Η ανησυχία πάντως που έχω και θέλω να μου πει πώς τα βλέπει ο Γενικός Διευθυντής είναι τι γίνεται με τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί εμείς στην Ευρώπη κάνουμε τεράστιες προσπάθειες σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Στον υπόλοιπο κόσμο όμως ακούμε λόγια, δηλώσεις καλών προθέσεων, αλλά δεν βλέπουμε να προχωράνε όπως προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε τελικά καταλαβαίνετε ότι η βιομηχανία μας έτσι μένει εφοπλισμένη, γιατί βλέπει ότι ο υπόλοιπο κόσμος δεν κάνει τα ίδια. Και με τις απειλές του νέου Προέδρου, του εκλογέτος Προέδρου των ΗΠΑ, όσον αφορά την τήρηση των συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί, μάλλον τη μη τήρηση. Καταλαβαίνετε ότι φοβόμαστε ότι δεν θα υπάρξει στήριξη. Λοιπόν, θέλω να ξέρω, Γενικός Διευθυντής, τι πιστεύει πρώτα απ' όλα για το πώς μπορούμε να πιέσουμε ώστε και ο υπόλοιπο κόσμος να κάνει όπως εμείς στα περιβαλλοντικά και πώς βλέπει τη συνέχεια τώρα που θα έχουμε νέο πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ο κύριος Μπράνερ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση που αφορά την αλλαγή του κλίματος. Κατά πόσο θεωρείτε ότι η πολιτική η οποία ουσιαστικά προχωρεί λίγο στο θέμα της απόδειξης για τις αλλαγές του κλίματος. Είναι κάτι που θα μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε ότι αυτά που κάνουμε σήμερα δεν θα είναι παροχημένα μετά από 10-15 χρόνια πριν ε, γίνω μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήμουν σε μια οργάνωση, την Christian Aid, για την αναπτυξιακή βοήθεια και βεβαίως το θέμα της αλλαγής του κλίματος που μας απασχολούσε σε μεγάλο βαθμό. Ένα τμήμα των ε, οργανώσεων στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας μας είχαν ε, επιστήσει την προσοχή στην αλλαγή του κλίματος και ότι αυτό βεβαίως είχε πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις για τους λιγότερο εύπορους ανθρώπους ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες και μάλιστα είχαμε ξεκινήσει και μία εκστρατεία με κεντρικό θέμα την ιστορία της φτώχειας. Αυτό που μας είχαν πει τότε πολλοί είναι ότι πραγματικά οι συνέπειες της αλλαγής του κλίματος είναι κάτι που βεβαίως πλήττει κατά κύριο λόγο τους φτωχούς. Σε κάθε ανα σώμενη χώρα βλέπουμε ότι περισσότεροι άνθρωποι πέφτουν στη φτώχεια και υποφέρουν από τη φτώχεια λόγω μεταξύ άλλων και της αλλαγής του κλίματος. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν που θα ήθελα να θέσω είναι το θέμα της απόδειξης για τις ε, κλιματικές αλλαγές είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε και το έχουμε στο κέντρο της πολιτικής μας. Το θέμα επίσης των δασών και της πολιτικής μας για θέματα δασών μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος. Μεταξύ βορρά και νότου ξέρουμε ότι υπάρχουν τρομερές ανισότητες στον τομέα αυτό της πολιτικής μας και τι κάνουμε για να επεκτείνουμε τα δάση αντί να τα καταστρέφουμε, πώς προστατεύουμε τις δασικές εκτάσεις, ιδιαίτερα σε κάποιες χώρες του κόσμου όπου αυτά τα οποία σήμερα προστατεύουμε και τα οποία συνεισφέρουν πολύ σημαντικά στην μείωση των ε, εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα πώς στηρίζουμε κάποιες καλλιέργειες, πώς προσπαθούμε να μειώσουμε τις ανισότητες στην πολιτική αυτή μεταξύ Νότου και Βορρά. Όσον αφορά λοιπόν την αλλαγή του κλίματος τα τελευταία 50 χρόνια, γνωρίζουμε πολύ περισσότερα και ξέρουμε ότι η πολιτική μας στον τομέα των δασών, στον τομέα της ε, καλλιέργειας και της παραγωγής, η χρήση λοιπασμάτων. που χρησιμοποιείται και στο βορρά και στο νότο θα πρέπει να γίνεται με συνετό τρόπο, με περιορισμένο τρόπο. Πρακτικές λοιπόν στον γεωργικό τομέα που συνεχίζονται εδώ και 50 και 100 χρόνια μπορεί να έχουν τεράστιες επιπτώσεις, πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην αλλαγή του κλίματος. Δεν το ξέραμε, σήμερα το ξέρουμε. Στην Ήπεθρο λοιπόν, στις αγροτικές ε, περιοχές πώς παρουσιάζουμε το θέμα της αλλαγής του κλίματος, το ρόλο της δασοκομείας και το ρόλο κάποιων συγκεκριμένων καλλιεργειών. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Γκέμπραντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Κρέσ που είναι σήμερα εδώ. Δεν θέλω να είμαι αγενής αλλά θα προτιμούσαμε να είχαμε τον ε, Επίτροπο Τίμερμαντς. Αυτός είναι επικεφαλής αυτού του προγράμματος πριν από ένα χρόνο, το Μάρτιο όταν ήταν εδώ. Είπε ότι αυτή η στόχη είναι εξαιρετικά σημαντική για να προωθήσει τους βασικούς και φιλόδοξους στόχους τους σαν επίτροπος, που είναι η αηφορία. Ιδού το αποτέλεσμα. Απογοητεύομαι ιδιαίτερα διαβάζοντας αυτά τα έγγραφα που μας υποβάλλατε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτον, γιατί αν συγκρίνουμε αυτούς τους στόχους με τους στόχους της χιλιετίας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι η αναγνώριση των Ηνωμένων Εθνών θέματα αηφορίας. Λέει ότι είναι προϋπόθεση για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια για να εξαλείψουμε τη φτώχεια. Χωρίς λοιπόν να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος, η καταπολέμηση της φτώχειας είναι ψευδέστηση. Προστασία των οικοσυστημάτων, τα άγρια είδη ζώων, το θέμα των αλλιευτικών πόρων, όλα αυτά, το οποία είναι τόσο σημαντικά για να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Οι στόχοι λοιπόν ε, αυτή της βιωσιμότητας θα έπρεπε να αναγνωρίζουν όλες αυτές τις ε, υποχρεώσεις και ανάγκες ε, καθώς και την πολιτική για μια καλύτερη ζωή στον πλανήτη μας. Ο Τίμερ μας λοιπόν υποσχέθηκε πολλά. Η Επιτροπή υποσχέθηκε πολλά και βλέπουμε ότι αυτοί οι στόχοι αν υλοποιηθούν, αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα όλων των πολιτικών μας. Ειλικρινά όμως, εδώ υπάρχει ένα εκτελεστικό απόσπασμα, μια εκτελεστική περίληψη θα έλεγα όλων αυτών που θα έπρεπε να προτείνει η Επιτροπή. Δεν βλέπω τίποτα παραπάνω, εκτός από την ομάδα των 20 επιτρόπων. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα μείνουν απ' έξω? Αυτό αναρωτιέμαι. Οκτώ. Οκτώ επίτροποι δεν ε, εμπλέκονται στο θέμα των στόχων. Τέλος αυτό είναι το αστείο κομμάτι. Δηλαδή δημιουργούμε ένα γραφειοκρατικό όργανο για άλλη μια φορά για να μην πάρουμε τις απαραίτητες πολιτικές αποφάσεις, για να μην κάνουμε τίποτα και αν πάρω το 14 και 15 στόχο, βιοπικιλότητα και ζωή στη γη και στην θάλασσα. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι κάτι θα κάνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή η οποία δεν μπορεί καν να αποφασίσει αν θα πρέπει να παραμείνουμε στην παρούσα νομοθεσία που αφορά την βιοπικιλότητα, την οδηγία δηλαδή για τα οικοσυστήματα. Στείλαμε μια επιστολή στο Γιούνκερ και η απάντηση ήταν απογοητευτική. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν εδώ η Επιτροπή, τι αρμοδιότητες έχει όταν μας λέει ότι θα αλλάξει η κατάσταση. Καθημερινά βλέπουμε ότι δεν κάνει τίποτα η Επιτροπή για θέματα αηφορίας. Το έβδομο σχέδιο δράσης για το περιβάλλον ήταν πολύ πιο φιλόδοξο από αυτά που βλέπουμε εδώ για τους στόχους. Και η Επιτροπή για την δράση σε θέματα κλίματος ήταν εξαιρετικά επικριτική από μέρους του ελεκτικού συνεδρίου. Δεν βλέπω λοιπόν τίποτα να αλλάζει στην καθημερινή μας δράση. Ο Φιλ Χόγκαν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σήμερα όταν τον ρώτησα για την αηφορία, τη βιωσιμότητα και τη γεωργία, μου είπε πρέπει να περιμένετε 7 χρόνια. Πραγματικά λοιπόν δεν βλέπω κανείς να βιάζεται, δεν βλέπω το θέμα να θεωρείται κατεπήγον και αυτό με απογοητεύει ιδιαίτερα. Πολύ συγκεκριμένα θα ήθελα να μιλήσω για τα κριτήρια βιωσιμότητας στο εξάμεινο. Αυτό όμως βλέπω ότι δεν συνεχίζεται από την παρούσα Επιτροπή. Αυτό βεβαίως συνάδει με τους στόχους αυτούς. Μήπως πρέπει λοιπόν να τους επαναφέρουμε. Επίσης η έκθεση του Κοινοβουλίου, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να αποτελέσει μια βάση, αλλά σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή θα πρέπει λιγάκι να ενδυναμώσει τις προσπαθίες της και το ρυθμό της για να συμμορφωθεί και με τα Ηνωμένα Έθνη πολύ σημαντικό να ακουστούν ε, όλες οι απόψεις των πολιτικών ομάδων. Έχετε το λόγο όμως και μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ και όλους τους ευρωβουλευτές. Η Επιτροπή εκτιμά όλους ιδιαίτερους να μπορούμε να έχουμε αυτήν την ε, πραγματική και ανοιχτή κουβέντα μεταξύ μας. Θα απαντήσω πρώτα απ' όλα στην κυρία Αγιούσο, η οποία είπε ότι στηρίζει την ανακοίνωση, ότι τους φάνηκε φιλόδοξη και ότι πιστεύει ότι η Επιτροπή αυτή μπορεί να είναι σύμμαχος της Κομισιόν. Ε, πράγματι. Και εμείς βασιζόμαστε σε εσά και ελπίζουμε ότι θα είσαστε μία από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές που θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση στο έργο μας υπέρ της επίτευξης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Ρωτήσατε πώς θα ενσωματωθεί σε όλα αυτά η επιχειρηματική κοινότητα. Μα τα βλέπει όλα αυτά σαν ένα όφελος, όχι σαν ένα εμπόδιο και αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που διαπιστώνουμε είναι ότι το περιβάλλον που μέχρι τώρα θεωρεί το εμπόδιο, σήμερα για τις επιχειρήσεις θεωρεί το όφελος γιατί επενδύουν στην βιωσιμότητα, γιατί θέλουν να αλλάξουν το μοντέλο τους το επιχειρηματικό και να το προσαρμόσουν στις ανάγκες του περιβάλλοντος. Άρα είναι πιο καινοτόμες επιχειρήσεις που έχουν και τα καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι είναι σημαντικό ο ιδιωτικό τομέα να συμμετέχει, όπω έγινε και με την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών. Εξού και ιδέα για αυτή την πλατφόρμα, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για να συνεχιστεί ο διάλογος, ώστε και ο ιδιωτικό τομέα να συμμετέχει. Και έτσι θα μπορούμε να έχουμε και ανταλλαγές απόψεις μαζί με τον ιδιωτικό τομέα για να δούμε ποιε είναι οι βέλτιστες πρακτικές στον κάθε κλάδο και με τη συμμετοχή βέβαια και των χωρών μελών. Αλλά με ρωτήσατε κάτι πολύ σημαντικό στο τέλος της παρέμβασής σας. Ρωτήσατε ποια είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ λοιπόν το πακέτο αυτό με τις τρεις ε, ανακοινώσεις πρώτη έχει να κάνει με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν και δύο ανακοινώσεις που καλύπτουν αυτό το ζήτημα. Η πρώτη είναι η πρόταση για μια νέα ευρωπαϊκή συνένεση όσον αφορά την αναπτυξιακή μας πολιτική. Στη πρόταση αυτή υπάρχει μια αλλαγή για την ατζέντα του 2030 και αυτή είναι η εταιρική σχέση. Πολλές φορές έχουμε κατηγορηθεί για πατερναλιστές. Αυτό που θέλουμε λοιπόν να κάνουμε τώρα είναι οι χώρες μέλη με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συνεργάζονται στα οριζόντια ζητήματα της αναπτυξιακής πολιτικής. Ε, βιώσιμη ενέργεια, κλιματική αλλαγή, επενδύσεις, μετανάστευση, κινητικότητα, ισότητα, θέματα που έχουν να κάνουν με την νεολαία γιατί θέλουμε να δώσουμε περισσότερη αξιοπιστία στην αναπτυξιακή μας πολιτική, να βασιστούμε σε κοινή ανάλυση, σε κοινή στρατηγική και σε ένα κοινό προγραμματισμό με τις υποανάπτυξη χώρες. Έτσι τίθεται το θέμα στη νέα συνένεση και ένα από τα σημαντικά εργαλεία μας είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Εξωτερικών Επενδύσεων με την δυνατότητα χρηματοδότησης ώστε να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη εκεί που περισσότερο χρειάζεται. Υπάρχει και η δεύτερη ανακοίνωση που μιλάει για μια νέα εταιρική σχέση με τις χώρες ΑΚΕ, τις χώρες Αφρικής, Καρυβικής και Ειρηνικού, εν ώψη του 2020. Η Ευρώπη είναι πολυμερής οργανισμός έτσι κι αλλιώς και ως τέτοιος πιστεύει ότι η συνολική και σφαιρική στόχη πρέπει να επιτεθούν πολυμερώς και να υπάρχει συμφωνία με τις χώρες ΑΚΕ, μια συμφωνία πλαίσιο, που να μπορεί να συμπεριλάβει και ειδικέ εταιρικέ σχέσεις για την Αφρική, για την Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Για τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών τώρα και τι θα γίνει μετά τις εκλογές στην Αμερική, Εκεί οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν συμφωνήσει με του αναπτυξιακούς στόχους. Οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δραστηριοποιηθούν ώστε να επιτεθούν αυτοί οι στόχοι και να κάνουν από μόνοι τους ό,τι πρέπει αλλά και να συνεργαστούν με τον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα, έρχομαι ε, στα ζητήματα που έθεσε ο κύριος ε, Γεβραντή. Πρώτον, πολύ σωστά Αναφερθήκατε στην κλιματική αλλαγή και είπατε, μα πώς η κλιματική αλλαγή θα διευκολυνθεί. Πρώτα απ' όλα, ένας από τους 7 ε, μάλλον ένας από τους στόχους, τους αναπτυξιακούς, ο αριθμός 13, είναι εκείνο που λέει να ληφθεί δράση για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Με αστερίσκο που λέει αναγνωρίζοντας ότι η Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή είναι και το κύριο διακυβερνητικό φόρουμ για να γίνουν διαπραγματεύσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι από τη μια πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τη Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή μετά τη Συμφωνία στο Παρίσι ιστορικής σημασίας και εκείνη του Μαρακές πρέπει να εφαρμόσουμε τους στόχους που συμφωνήθηκαν αλλά επιπλέον σημαίνει ότι πρέπει την κλιματική αλλαγή να τη λάβουμε υπόψη μας σε όλες μας τις πολιτικές. Συνεπώς, η κλιματική αλλαγή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να ενταχθεί στις πολιτικές μας και το κάνουμε αυτό με τα για του θερμοκηπίου, για την ενεργειακή απόδοση, αλλά επιπλέον πρέπει να αφιερώσουμε τουλάχιστον 20% του ευρωπαϊκού προπολογισμού σε δράσεις για το κλίμα. Όλα αυτά έχουν συμφωνηθεί και πρέπει σιγά σιγά να εφαρμοστούν. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που νομίζω θα σας ενδιαφέρει. Τι θα κάνουμε με τις αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί μερικές αντιμετωπίζουν τραγικές καταστάσεις εξαιτία της κλιματικής αλλαγής. Με τη Συμφωνία των Παρισίων ξέρετε ότι υπάρχει η δέσμευση για 100 δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να κινητοποιηθεί χρηματοδότηση και έχουμε και άλλα στοιχεία υπέρ του κλίματος. Θα ασχοληθούμε για παράδειγμα με τη δασοκομεία. Η δασοκομεία η συμπεριλαμβάνεται στο στόχο 15 που καταπολεμά την αποψήλωση αλλά προωθεί οικοσυστήματα και επιβραδύνει την απώλεια βιοποικιλότητας και μιλάει και για διαχείριση, ε, βιώσιμη διαχείριση των δασών. Άρα, στη στρατηγική μας για την ε, βιοποικιλομορφία, που έχει πολύ φιλόδοξο στόχο να επιβραδύνει την επιδείνωση μέχρι το 2020. Αυτό σημαίνει ότι, στη βιωσιμότητα, η βιωσιμότητα στη διαχείριση των δασών θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Πρέπει λοιπόν να έχουμε απάντηση στο στόχο 15. Άρα σας διαβεβαιώνω και τονίζω ότι τα τρία θέματα στα οποία αναφερθήκατε καλύπτονται απόλυτα στη στρατηγική. Τώρα, στη συνέχεια, ε, ο κ. Κυπραντή δεν ήταν πολύ ευτυχισμένος από την ανακοίνωση. Ε, ζητώ συγγνώμη που δεν είναι εδώ ο κύριος Τίμερμανς. Ε, πρέπει να κάνετε με μένα. Σίγουρα λυπάτε που δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί σας. Αλλά να ξέρετε ότι παρά το γεγονό ότι δεν μπορούσε να έρθει εδώ σήμερα, θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντική η επιτροπή σας και τα θέματά της και να ξέρετε ότι κάνει ό,τι μπορεί στην Επιτροπή πέρα αυτών. Τώρα η βιωσιμότητα είναι ζωτική σημασίας για να απαλληφθεί φτώχεια. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να μεταφέρουμε πιο πέρα. Η βιοπικιλότητα, το νερό, η αγρία ζωή, όλα αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα παίρνει πολύ στα σοβαρά. Θα είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι από αυτό το Σαββατοκύριακο στο Καλκούν στην διάσκεψη κόπη για την βιοπικιλότητα. Όλοι μιλάνε για την κλιματική αλλαγή, αλλά υπάρχει και άλλη όψη του νομίσματος που είναι η Σύμβαση για την Βιοπικιλότητα. Έχουμε λοιπόν μια πολύ σημαντική ε, συνδιάσκεψη τους επόμενους μήνες και πρέπει να ληφθεί δράση για την προστασία της βιοπικιλότητας. Σας διαβεβαιώνω και σας ευχαριστώ γιατί συνεργαστήκατε μαζί μας και στο ΣΑΠΣ και τα είδατε κι εσείς με τα ίδια σας τα μάτια τι γίνεται για την άγρια ζωή. Εδώ έχει ληφθεί δράση. Λέτε ότι πρόκειται για μία περίληψη. Κατά κάποιο τρόπο έχετε δίκιο. Η ανακοίνωση αυτή είναι ένα σημείο εκκίνησης. Ποιες είναι οι πολιτικές και πώς συνδέονται μεταξύ τους οι 17 στόχοι και πώς συνδέονται με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό είναι κάτι επιπλέον. Η πολιτική εφαρμογή όμως των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο έγγραφο αυτό, το οποίο εντοπίζει τους στόχους, δίνει μια φωτογραφία, αν θέλετε, το που βρισκόμαστε τώρα και λέει τι θέλουμε να πετύχουμε. Πριν σας μίλησε για τους στόχους του 14 και 15. Υπάρχει και το Natura 2000. Στην επόμενη εβδομάδα στο Σώμα των Επιτρόπων θα συζητήσουμε για τις οδηγίες όσον αφορά το Natura 2000. Θα υπάρξει κάποια συνομιλία Σούλτς Γιούγκερ για προσανατολισμούς και στη συνέχεια θα υπάρξουν ειδικέ ανακοινώσεις για τις αντικές όσον αφορά την βιοποικιλομορφία και εδώ πρέπει να εφαρμόσουμε κάποια στρατηγική θα έχουμε και την ανακοίνωση για το ενεργειακό που θα συμμετέχουν διάφορες γενικές διευθύνσεις και για την κλιματική αλλαγή και για την ε, πρόσβαση σε πόρους κτλ. Λοιπόν, σε αυτό το έγγραφο μιλάμε για τους στόχους χωρίς να παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις για τον καθένα από αυτόν. Απαριθμίζουμε το τι πρέπει να κάνουμε και από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να δουλεύει είτε με την Ενεργειακή Ένωση, είτε με την παρελθοντική πολιτική, είτε με την κυκλική οικονομία κλπ. κλπ. Πρέπει επίσης να δούμε και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Πώς θα καλύψει το δικό του ρόλο, θα φέρει σε πέρα το δικό του ρόλο. Και γι' αυτό εδώ πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δούμε ποιες είναι οι θέσεις μας. Υπάρχει και η διαδικασία του εξαμήνου. Ρωτήσατε, η βιωσιμότητα θα είναι κριτήριο μέσα στη διαδικασία του εξαμήνου. Κατά τη γνώμη μας, μετά από την έγκριση των 23 στόχων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις πολιτικές και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να πούμε ότι θα κάνουμε πρόοδο. Οπότε, για τα σχόλια του κ. Γκεμπραντή θα πω ότι ναι, μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την ανακοίνωση, επειδή είπατε εσείς ότι δεν τη βλέπετε αρκετή δυνατή, στην εφαρμογή θα φανεί. Επί της ουσίας πιστεύω ότι έχουμε υψηλού επίπεδου φιλοδοξίες. Είναι η πιο σημαντική πρόκληση και δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας που συμφώνησαν για τα επόμενα χρόνια. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας, περιβάλλοντος. Έχουμε και την δυνατότητα να βελτιώσουμε τα στοιχεία της ανακοίνωσης και από εκεί πέρα να δούμε και τα στοιχεία της διαδικασίας, γιατί και η διαδικασία πρέπει να είναι καλή ώστε να ε, υπάρχει συνοχή, να διασφαλίζεται συνοχή. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις, την έκθεση πρωτοβουλίας και φυσικά πολύ θα θέλαμε η δικιά σας επιτροπή να συνεργαστεί και με τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές που και αυτές θα είναι ιδιαίτερα δραστήριες για την επίτευξη των στόχων ε, της βιώσιμης ανάπτυξης. Υποσχέθηκα στους ε, επιτρόπους ότι θα σας πω και ίσως έρθει και ο κύριος Τίμερμανς. Και έτσι να έχουμε όλους τους επιτρόπους και τους 28. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας και νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας συνεδρίαση. Ξεκινήσαμε στις 9 σήμερα το πρωί με τους συντονιστές και θα ξανασυναντηθούμε στις 8 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ.